Κυρίε Κυρίες και κύριοι, άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας προβλέπει δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16 Σεπτεμβρίου 2010. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Εργμάν Βαν Ρόμπεϊ. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δίνουμε αμέσω το λόγο. Παρακαλώ κύριε πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16 Σεπτεμβρίου 2010 συνεκλήθη κατά κύριο λόγο για να εστιάσει στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και μια μικρή προγραμματισμένη συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματο για την ομάδα εργασίας ε, για την οικονομική διακυβέρνηση και μια εκτό προγράμματο συζήτηση για την κατάσταση των Ρωμά. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε όλα αυτά τα θέματα με τη σειρά. Πρώτον, για τα εξωτερικά ζητήματα. Πριν από 8 μήνε όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου και επισκέφθηκα τι πρωτεύουσε, ε, διαπίστωσα μια απογοήτευση μετά τη σύνοδο Κορυφή τη Κοπενχάγη. Ε, και υπήρχε η αίσθηση ότι ήταν παραγωνισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οικονομικά ήταν ζωφερά, ενώ άλλε περιοχές του κόσμου αναπτύσσονται ε, με οικοργούς ρυθμούς. Επιπλέον αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη ορισμένων κρατών γίνεται ουσιαστική πολιτική ισχύς. Το G20 ενώ ε, ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προβληματικό για την Ευρώπη όπως και η εκπροσώπησή της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμφανίζονται νέοι ε, πρωταγωνιστές ε, πλέον και η συνθήκη της Λισαβόνας ε, απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσει τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσει στρατηγική καθοδήγηση στις εργασίες των άλλων θεσμικών οργάνων. Χαίρομαι που όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν να προσιλωθούν στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν ε, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εστερνιστεί περισσότερο αυτά τα θέματα και να λάβουν τις ευθύνες τους εκείνοι ε, ως μέλη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης αυτής. Τι συζητήσαμε τώρα. Φαίνεται επίγον για μένα να ασχοληθούμε πρώτα με τις στρατηγικές μας εταιρικές σχέσεις συγκεκριμένους στόχους ε, και συγκεκριμένα έργα στην πράξη πρέπει να ε, ορίσουμε. Πώς καλύτερα θα αξιοποιήσουμε τις συνθήκη Λισαβόνας με τη νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο ε, ε, για ε, τη συμφωνία του σε αυτό το θέμα. Πώς θα βεβαιωθούμε ότι όσα γίνονται από τις Βρυξέλλες και τις πρωτεύουσες πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Πώς μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα τους διαφόρους ε, πρωταγωνιστές της Βρυξέλλες. Πώς θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με εταίρους κατά τη διάρκεια συνόδων κορυφής σε τομείς όπως είναι η οικονομία, η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια. πώς ε, αντιμετωπίζουμε τους εταίρους έναν ένα. Έχουμε προτεραιότητες λοιπόν τώρα θέση σε συγκεκριμένα θέματα. Και οι βασικές μας αρχές και τα μηνύματα προς τρίτε χώρες της Συνόδου Κορυφή θα πρέπει να ε, βασίζονται σε κειμένε διαπραγματεύσεις και ε, ανταλλάγματα. Πρώτον, ε, Ω προ τη διαδικασία αυτή πρέπει να πούμε ότι είναι η αρχή τη διαδικασία. Και δεύτερον, τα βασικά μα μηνύματα θα πρέπει να είναι αντικείμενο εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να, ε, ε, να ετοιμάζει και να τα εκπονεί το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, η ΥΠΑΤΗ Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Όπω προετοιμάζουμε και ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη συνεδριάση του G20. Τρίτον, με του εταίρους μα, βασική έννοια είναι η αμοιβαιότητα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε και η ταυτοποίηση ε, κοινών ε, μηβαίων συμφερόντων. Ε, υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι αυτό ακόμα δεν συμβαίνει. Θα επιμένουμε σε στόχους που πρέπει να γίνονται πραγματικότητα, πάντα συγκεκριμένα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε αγαπητοί συνάδελφοι και περισσότερο μια στρατηγική Έχουμε ιδέες συζητήσει και αναπτύξει πώς θα τοποθετηθούμε απέναντι στην Κίνα, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη επεξεργασία αυτό. Όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ συναντήσαμε θα συναντήσουμε συγγνώμη, τον Κινέζο Πρωθυπουργό, δεν θα μιλήσουμε μόνο εξ ονόματο των Βρυξελών, αλλά και των 27 κρατών μελών. Ασχοληθήκαμε και με άλλε επικείμενε συναντήσει. Η Σύνοδο Κορυφή του G20 στη Σεούλ και ε, ε, άλλη σημαντική σύνοδος επίκυνται το Νοέμβριο. Θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε στις 28 και 29 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, τις ε, προτάσεις μας αυτές. Η Γαλλία που αναλαμβάνει την Προεδρία το 2011 έκανε προτάσεις και ο Γάλλος Πρόεδρος συγκεκριμένα για να δώσουμε μια νέα δυναμική στο G20 και να είναι μια ολόκληρη διαδικασία ε, η Σύνοδος Κορυφής και όχι απλώς μια διοργάνωση, ένα γεγονός. Στη Μέση Ανατολή είναι στρατηγικό συμφέρον να πετύχουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης. Ειδική ανακοίνωση εγκρίναμε σε σχέση μάλλον με ε, την κοινή θέση του Δεκεμβρίου 2009, συμμετέχουμε μέσω της τετραμερούς στη διαδικασία αυτή. Τα Δυτικά Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή τους προοπτική μας απασχόλησαν επίσης και η ανατολική εταιρική σχέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η φήμη μας στον κόσμο αρχίζει από τη σταθερότητα στην ίδια μας την Ήπειρο. Αν θέλει κανείς να είναι πρωταγωνιστής παγκοσμίω, θα πρέπει να είναι περιφερειακή δύναμη πρώτα απ' όλα. Από τώρα και στο εξή θα συζητούμε υπό αυτό το πνεύμα την εξωτερική πολιτική στο Συμβούλιο. Μόνο έτσι θα είμαστε ε, αξιόπιστοι και ισχυροί, αν είμαστε ενωμένοι. Δείξαμε την ενότητά μας στη θέση των 27 για επιπλέον κυρώσεις για το Ιράν που δεν ήταν προφανές αυτό. Και επίσης ε, πολύ σημαντικό ψήφισμα του για το διάλογο μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Άλλο πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο θέμα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκτός από τη στρατηγική αυτή και τη συζήτηση γενικά, ε, καταλήξαμε και συμπεράσματα για δύο συγκεκριμένα θέματα, την Νότια Κορέα και το Πακιστάν. Εκεί φάνηκε απολύτως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είναι ενωμένη μπορεί να έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ε, συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Νότια Κορέα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα εξωτερικής πολιτικής. Αφορά τη ζωτική σχέση ε, με μια πολύ μεγάλη εμπορική χώρα, αλλά όχι μόνο αυτό, και για το σύνολο της ασιατικής οικονομίας. Ε, επί μια τριετία είχαμε φτάσει κοντά στη συμφωνία και τώρα είναι γεγονός. 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα ε, κερδίσουν οι Ευρωπαίοι και συγκεκριμένα εξαγωγική βιομηχανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την απασχόληση και για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Για το Πακιστάν θέλουμε να υποστηρίξουμε ε, τα μάλα τη χώρα αυτή αφού επλήγει τόσο ικτρά από τις καταστροφικές πλημμύρες. Περισσότερη βοήθεια και περισσότερο εμπόριο. Θέλουμε το Πακιστάν τώρα να ε, ανακτήσει και να αναπτυχθεί οικονομικά. Η κάθε Άστον μας βοήθησε να συμφωνήσουμε και για αυτό το σημαντικό θέμα και για μεγαλύτερη πρόσβασή του στην αγορά. Ένα δεύτερο σημείο τώρα. Η ομάδα εργασία, Task Force, κατά τη ε, διάρκεια του γεύματο, συζητήσαμε για την οικονομία, για το πώς ε, θα προχωρήσουμε πολιτικά. Στο πρώτο εξάμεινο ε, του ε, τρέχοντος έτους ασχοληθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με επίγοντα οικονομικά θέματα. Είναι κάπως καλύτερα τώρα οι οικονομίες μας, αλλά δεν έχει περάσει η κρίση ακόμα. Κατά τη διάρκεια ε, του γεύματος ενημέρωσα τους συναδέλφους για την οικονομική διακυβέρνηση και χθε στο κοινοβούλιο σας οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιθυμούν να συνεχίσουν ε, την εργασία αυτή και να διατηρήσουν την ορμή που έχει αναπτυχθεί. Έχουμε μεγάλη ε, συνένεση επιτύχει για σημαντικά θέματα όπως είναι η μακροοικονομική εποπτεία και το αντίστοιχο πλαίσιο για να παρακολουθεί την κατάσταση και να διορθώνει κάποιες αδυναμίες, κάποιες ανισορροπίες. Επίσης, συμφωνία για ενίσχυση των εθνικών δημοσίων οικονομικών και να μεταφέρεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία πραγματικά ε, στην ε, εθνική νομοθεσία. Επίσης αποφασίσαμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Επίσης ε, προχωρήσαμε και στο θέμα των κυρώσεων με επτά προέδρους επιτροπών σας και αρχηγούς πολιτικών ομάδων εχθές είχαμε μία συνεδρίαση και τα εξήγησε αυτά και πώς θα ενισχυθεί ο οικονομικός πυλώνας της ΟΝΕ. Ορισμένοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους ότι προχωρούν με αργούς ρυθμούς αυτά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η πρόοδος που έχει γίνει. Σε σχέση με το 1997 για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το 2005 στην αναθεώρησή του, οι ρυθμοί που ακολουθούμε σήμερα είναι πολύ πιο γρήγοροι παρά ε, το περίπλοκο των θεμάτων. Το Σεπτέμβριο, στις 27 του μηνός, θα ολοκληρώσουμε στην Task Force και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Οκτωβρίου και στις 28 και 29 Οκτωβρίου θα μπορεί να λάβει απόφαση το Συμβούλιο. Νομοθετική πρόταση προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί τα τέλη Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την νομοθετική της ε, πρωτοβουλία, προτάσεις που θα έρθουν στο Κοινοβούλιο σα βεβαίως προς συζήτηση και έγκριση με τις ε, νομοθετικές διαδικασίες θετικά μπορούν να συμβάλλουν οι προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εξελίξης. Κερδίσαμε τη μάχη του ευρώ και ε, τον άλλο μήνα πραγματικά πιστεύω θα βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα για την κρίση. Τρίτο θέμα, η Ρωμά. Κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήσαμε αυτό το θέμα που σας ενδιαφέρει πολύ. Συνένεση επιτεύθηκε για πέντε ζητήματα, αλλά δεν εκφράστηκε αυτό ως ε, επίσημο συμπέρασμα του Συμβουλίου. Πρώτον, ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα και το καθήκον να αναλαμβάνει δράση για να διατηρεί το κράτος δικαίου στην επικράτειά του. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να βεβαιώνει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς το κοινοτικό δίκαιο και έχει και δικαίωμα και καθήκον να κάνει έρευνα σχετικά. Τρίτον, σημειώσαμε τη δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τέταρτον, σεβασμός είναι ο βασικός κανόνας της σχέσης μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πέμπτον, σε μελλοντική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συζητήσουμε το θέμα της ένταξης των Ρωμά. Απαγορεύεται κάθε είδου διάκριση που να βασίζεται στο φύλλο, στην εθνότητα ή στην εθνικότητα. Είναι θεμελιώδη αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σεβασμό τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι από τι βασικότερε αξίε μα και αρχές μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να θεωρούνται πάντα σύνοδοι κορυφή, αλλά συνεδριάσεις ρουτίνα σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεδριάζει ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Επιτρέψτε μου να τονίσω εδώ ότι τώρα που γίνεται νέα συζήτηση για κοινοτικά θέματα στο κοινοβούλιο σα, πρέπει να σα θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι θεσμικό όργανο. Ε, και συνεδριάζει και στο G8 και στο G20, είναι θεσμικό όργανο πλέον της Ένωσης και ε, καθοδηγεί και τα κράτη-μέλη σε από υψηλό επίπεδο πολιτικό και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι συμμετέχουν στα κοινοτικά πράγματα γιατί έτσι μόνο θα επιτύχουμε. Εκεί δεν συμμετέχουν μόνο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα ότι εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικών. Συχνά δε παρευρίσκεται και ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις συνθήκες Λισαβόνας και μετά προεδρεύεται από κάποιον ε, που δεν εκπροσωπεί ταυτόχρονα και ένα κράτος μέλος, αλλά θα πρέπει να εργάζεται και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και σε στενή συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα για να ζητεί λύσεις υπέρ του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Γι' αυτό το λόγο επενδύω και χρόνο και ενέργεια για να διατηρώ τακτικές επαφές με τους προέδρους των άλλων θεσμικών οργάνων, τουλάχιστον τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ε, Περιτροπή ε, Προεδρία του Συμβουλίου, την Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωζώνη, το Eurogroup και σας, βεβαίως κύριε Πρόεδρε μαζί με Προέδρους ε, πολιτικών ομάδων και κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πολύ πέρα από τα όσα ορίζει η συνθήκη λοιπόν. Εργαζόμαστε πραγματικά υπέρ του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Καταβάλλονται προσπάθειες από όλα τα θεσμικά όργανα. Και τους τελευταίους μήνες ε, είδαμε ότι αυτές οι ε, προσπάθειες έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς. Οι οικονομίες μας ε, ανατάσσονται ελπιδοφόρα και σιγά σιγά επανέρχεται και η εμπιστοσύνη με την νομοθετική προσπάθεια στα θέματα εποπτείας. Και πολλά κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, έχουν λάβει με μέτρα θάραλέα σε πολύ δύσκολες πολιτικές ε, περιστάσεις. Σε περισσότερα, τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη δεν έχει παρέλθει η κρίση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απασχόληση, παρόλο που υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις. Τώρα είμαστε σε καλύτερη μοίρα από ότι στο παρελθόν. Χρειάζεται όμως και απομένει πολλή δουλειά να γίνει. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα την κάνουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, ομιλία σας ε, και τις παρατηρήσεις σας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Ο Αντιπρόεδρος Μάρος Σέτσκοβιτς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Κοινοβούλιο υπήρξε πάντοτε σαφές ότι από τα βασικότερους στόχους της συνθήκης της Λισαβόνας είναι να ισχυροποιηθούμε ε, στη διεθνή ε, σκηνή. Προσπαθούμε να ε, μεγιστοποιήσουμε τις φωνές μας στον κόσμο ούτως ώστε να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας και τις αξίες μας και να συμβάλλουμε στις παγκόσμιες προσπάθειες απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις, κλιματική αλλαγή, έλλειψη πόρων, η οικονομική κρίση. Έχουμε ευκαιρίες και έχουμε και ευθύνε. και η συνθήκη της Λισαβόνας μας έδωσε τα εργαλεία να επιτύχουμε τους στόχους μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, συνεχίζεται όλη η εργασία Πρέπει στις χώρες μας να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Με τους εταίρους μας πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιστικός συνομιλητής. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά νομίζω ότι ήταν βασικό βήμα προόδου η Σύνοδος Κορυφής. Στους εννέα μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Η Βαρόνι Άστον ε, τώρα είναι η φωνή της Ευρώπης στη διεθνή κονίστρα και με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου ελπίζω να έχουμε σύντομα ε, την, ε, υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εν λειτουργία. Έχει, έχουν αναλυφθεί ε, λειτουργίες για εκπροσώπηση και συντονισμό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδιορίσε τα επόμενα βήματα τόσο ως προς τη μορφή όσο ως προς την ουσία. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έχουμε μια πιο συνεκτική πολιτική απέναντι στους στρατηγικούς εταίρους, κυρίως ως προς την Κίνα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανήλθε στην προσπάθεια ε, μιας κοινή ε, προσέγγισης. Ξέρουμε μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ε, έχουμε πρέπει να πούμε στους εταίρους μας ότι, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε για αυτό το οποίο θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρχουν διστάμενες απόψεις μεταξύ των κρατών μελών, διότι υπονομεύουν αυτό το μήνυμα. Ο πρόεδρος Βαρομπέ και ο πρόεδρος Μπαρόζο μιλούν, μίλησαν στο Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μιλώντας για ένα πραγματικό κονσένσους, ε, για μια κοινή δέσμευση, για μια κοινή ατζέντα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ήταν σημαντικό να προσδιορίσουμε ειδικά συμφέροντα απέναντι στους στρατηγικούς μας εταίρους και να μπορέσουμε να εκπέμψουμε το ίδιο μήνυμα παγκοσμίω προς τους εταίρους μας. Πρέπει ε, να ασχοληθούμε με την Κίνα, Ινδία, Ρωσία και, οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε το φθινόπωρο και με το G20 το Ευρωασιατικό ε, Συνέδριο και επίσης το Αφρικανικό Συμβούλιο Κορυφής αναγνωρίστηκε το εμπόριο ως βασικό θέμα. Είναι ένα σύμβολο ισχυρό ότι πρέπει να έχουμε συμφωνία με την Κορέα. Και αυτό μας δείχνει ότι είναι φυκτό. Αυτά ε, ήταν μια συμφωνία που συνάφθηκε που δεν ήταν εύκολη αλλά οποία εμπεριέχει ευκαιρίες ε, μεγάλων ε, πλεονεκτημάτων και κερδών. Πρέπει να βοηθήσουμε βεβαίως το Πακιστάν. Ήδη κάνουμε πολλά με ανθρωπιστική βοήθεια και με ανακτυψιακή βοήθεια πράγμα που θα είναι κρίσιμη για την ανοικοδόμηση αυτής της χώρας. Αλλά θα έπρεπε να πούμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την μακροπρόθεσμη προοπτική της ανάπτυξης του Πακιστάν διαμέσου εμπορικών ε, μέτρων. Θα γίνουν προτάσεις ε, τον επόμενο μήνα. Η Προεδρία του G20 από την Γαλλία θα είναι μια καλή ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα έχουν προτεραιότητα ευρωπαϊκή στόχη. Η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει αυτό το φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα έτη. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για δύο άλλα θέματα. Οικονομική διακυβέρνηση, οι εργασίε Τη της ειδική ομάδας είχαν ως πρόεδρο τον κύριο Φαντρομπό και έγιναν προτάσεις από την Κομισιόν και δείχνουν ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά από το Μάιο. Η Επιτροπή θα υποβάλει την επόμενη εβδομάδα προτάσεις και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή ε, για την φάση συναπόφασης για να μπορέσουμε να εξετάσουμε νομοθετικές προτάσεις εν ώψη του νέου συστήματος που θα πρέπει να εγκατασταθεί στα μέσα του επομένου έτους. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να αρχίσουμε γρήγορα να εξετάζουμε αυτές τις προτάσεις. Το πακέτο θα έχει τρεις στόχους. Πρώτα απ' όλα να ενισχύσουμε την συμμόρφωση των κρατών στο Σύμφωνο σταθερότητας να διευρύνουμε την οικονομική εποπτεία για να μην υπάρχουν ανισορροπίες και η οικονομική εποπτεία να έχει κίνητρα για συμμόρφωση ε, προοδευτικά που να εφαρμόζονται δίκαια και να μπορούν να είναι αποτελεσματικά αυτό οδηγεί σε μεγάλη ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής μας διακυβέρνησης, κυρίως για την Ευρωζώνη. Αυτή η ατζέντα θα εμβαθυνθεί ακόμα περισσότερο όταν η ειδική ομάδα κάνει την τελική της έκθεση τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Κορυφής. Και τέλος το θέμα των Ρωμά. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω ένα σημείο. Η Επιτροπή έχει εδώ ευθύνη ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Και Είμαστε αρκετά σαφείς σχετικά με τις ευθύνες μας δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο και θα υπερασπιστούμε ε, τις, ε, τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Θα δούμε λοιπόν αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει τηρηθεί και ε, ως προς τα μέτρα κατά των διακρίσεων. Θα κάνουμε αναλύσεις και σύντομα το Κολέγιο των Επιτρόπων θα εξετάσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε αυτό που το ουσιαστικό μέρος αυτής της συζήτησης που είναι να ελαφρύνουμε το βάρος στην οδύνη των Ρωμά και να επιτρέψουμε καλύτερη ενσωμάτωση. Παράλληλα λοιπόν εξετάζουμε πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις προτάσεις του Απριλίου για με, ούτως ώστε με τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να επιτρέψουμε καλύτερη ενσωμάτωση των Ρωμά. Έχουμε μια ειδική ομάδα για να δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε απτά μέτρα για την ενσωμάτωση και η Task Force θα συναντηθεί για πρώτη φορά σήμερα το πρωί και ε, στο τέλος αυτού του έτους θα υποβάλει τα της και ξέρω ότι το Κοινοβούλιο αυτό θέλει να ενημερώνεται ε, τακτικά για τις προόδους των εργασιών αυτών και η Κομισιόν θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Εν κατακλείδη συζητήσαμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ικανότητα ε, δράσεως που έχουμε εσωτερικά και εξωτερικά για καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όργανα εργάζονται εντατικά και η Κομισιόν περιμένει καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο αυτό, να εμβαθύνει σε αυτήν την συνεργασία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις πολιτικές μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο πρόεδρος Τζόζεφ Ντόλ από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε Μπουζέκ, κύριε Βαν κύριε Σέρκοβιτ, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε τη σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με του διεθνεί εταίρου τη και την ε, χρηματοπιστωτική εποπτεία. Όμω το κοινό έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συζήτηση σχετικά με του Ρωμά. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω τη θέση τη ομάδα μου στο εξή. Κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να σέβεται τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τα όσα ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων, η οποία θα πρέπει να τα διασφαλίζει βεβαίω με τη μεγαλύτερη αμεροληψία. Όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι ισότιμα εναντί τη νομοθεσία και αυτό καθορίζει την ε, ισχύ τη Ευρώπη. Έτσι λοιπόν σεβόμαστε την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει διευκρινήσει από τη Γαλλία για τα μέτρα που έλαβε και δεν αμφισβητούμε ότι η Γαλλία θα απαντήσει πολύ σύντομα σε αυτό το αίτημα. Έπειτα η ομάδα του ΕΛΚ λυπάται για τα δυσάρεστα επεισόδια που συνέβησαν ε, στο πλαίσιο αυτό και ελπίζει ότι οι αξίες ε, της αλληλεγγύης και του σεβασμού του ανθρώπου, της ειρήνης και του αμοιβαίου σεβασμού ε, θα συνεχίσουν να είναι ένας κανόνας συμπεριφοράς για τις σχέσεις μεταξύ κρατομελών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τέλος, η ομάδα μου θυμίζει ξανά ότι ο ορισμός, ο καθορισμός και η υλοποίηση ευρωπαϊκών κοινών λύσεων για την ενσωμάτωση όλων των ε, μειονοτήτων στην Ευρώπη κατά την σημερινή κρίση είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι δημιουργούνται καταστάσεις ε, δυσαρέσκειας στις σχέσεις των μειονοτήτων με τις πληθυσμούς των χωρών υποδοχής. Θα πρέπει, κυρίε και κύριοι, κάθε πολίτης να μπορεί να απολαμβάνει των δικαιωμάτων του, αλλά καθένας να συμβαδίζει και με τις υποχρεώσει που ανταποκρίνονται στα δικαιώματα αυτά. Βεβαίως η ένταξη των ε, πολιτών είναι ένα δικαίωμα. Όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει σκοπό να κάνει καμία παραχώρηση και θα πρέπει ο νόμος να γίνεται σε κάθε περίπτωση σεβαστός. Η ένταξη στη χώρα υποδοχής, η εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, ο σεβασμός της διοκτησίας ε, των άλλων είναι δικαιώματα των οποίων ε, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ε, ισχύ. Αυτή είναι η τοποθέτηση της ομάδας μας. Μία ομάδα που βασίζεται σε κοινέ αξίες και ξεπερνά την ιδεολογία μιας μόνο παράταξης. Κάτι που φαίνεται ότι υπήρξε παγίδα για κάποιου τι τελευταίε ημέρε. Και επίση θα ήθελα να θίξω και άλλα δύο σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή, τη θέση μα στο Διεθνέ Προσκήνιο και την χρηματοπιστωτική εποπτεία. Ε, για το πρώτο θέμα, το θέμα που τίθεται είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε σεβασμό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πρωτοπόρος ε, στο διεθνές προσκήνιο και ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα φανήκαμε απόντε όμως το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Παλαιστίνη. Ε, κύριε Πρόεδρε, φροντίστε αυτό να αλλάξει. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρουν και δίνουν ενδιαφέρουσες ιδέες για το ποιοτικό άλμα που θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει ως πολιτική δύναμη να βαρύνουμε ως ενιαία δύναμη, όχι με 27 αντικρουόμενες διπλωματικές δυνάμεις. Για αυτή την ένωση, κύριε Πρόεδρε, σε εσά υπολογίζουμε. Είναι θέμα απόφαση και μεθόδου να αναγνωριστεί και να γίνει σεβαστή η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Επίση, οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να εξορθολογιστούν και η υπηρεσία εξωτερική δράση θα πρέπει να κάνει τα πρώτα βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Σκέφτομαι επίση ποια είναι τα κονδύλια που διαθέτουμε, ιδίω στον τομέα τη ασφάλεια και τη άμενα, τα οποία θα πρέπει να δαπανώνται με σωστότερο, ορθότερο τρόπο και με κοινέ μεθόδου. Απέχουμε ακόμη από αυτού του κοινού στόχου, όμω ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν του ερχόμενου μήνε έστω και μερικού από του στόχου που αναφέροντα τα συμπεράσματά σα. Για την οικονομική διακυβέρνηση τώρα, πρέπει να πω ότι η ομάδα μου είναι υπέρ των ε, πρώτων ε, λύσεων που πρότεινε η ομάδα εργασία Φαν Ρομπέι, ιδίω ε, για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητα με αυτερότερε κυρώσει. Θα πρέπει λοιπόν στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και τι αυταπάτε που είχαμε αναπτύξει τόσα χρόνια να δούμε ότι η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι μόνο μέσω τη οικονομική διακυβέρνηση και τη κοινωνική ορθή διακυβέρνηση όμω. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτ από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Κύριε Φαν σας άκουσα προσεκτικά και τη σύνοψή σας και την ομιλία σας. Όλα καλά στο Συμβούλιο, κανένα πρόβλημα. Ε, παραδέχομαι ότι εσείς ήσασταν παρόν, εγώ όχι. Ε, ζήσατε διαζώσει τη συζητήση εκεί, εγώ όχι. Παρ' όλα αυτά κάπω διαφορετικά αντελήφθην εγώ ε, το τι έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από αυτά που μας είπατε εσείς σήμερα. Τι ζήσαμε, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις. Οι ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, στράφηκαν κατά της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Τέσσερις ελευθερίες από το Μαστρίχτ έχουμε εγγυημένες. Ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εμπορευμάτων, του κεφαλαίου, των επιρρησιών και των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων θα πρέπει ακόμα να αποκτήσει ε, την ίδια ισχύ με την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου στην Ευρώπη. Και Καμιά φορά εύχομαι να είμαστε εξίσου επιμελείς ε, στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων με την αντιμετώπιση που έχουμε στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Τι ζούμε. Εσείς το υπενηχθήκατε αλλά δεν το εξηγήσατε. Σε αυτή την εποχή μετά τη Λισαβόνα που διανύουμε τώρα, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αγωνιστούν για να αναλάβουν τη θέση τους, τη θεσμική κάθε φορά. Και το νέο αυτό θεσμικό όργανο που εκπροσωπείται από εσά και είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρχηγών και κυβερνήσεων, γιατί από τη Λισαβόνα μόνο και μετά έχει γίνει θεσμικό όργανο. Προσπαθεί λοιπόν αυτό το θεσμικό όργανο να κατοχυρώσει τη θεσμική του ισχύ. Αυτό δεν είναι αθέμητο, το κάνει κάθε άλλο θεσμικό όργανο. Αλλά σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν εντό του Συμβουλίου υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Στη διαδικασία αυτή μετά τη Λισαβόνα έχουν εκχωρηθεί ε, αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κοινοτική λοιπόν διάσταση και το προβλέπει η συνθήκη. Ε, όλα αυτά ε, κινδυνεύουν να πέσουν ε, στην διάκριση, στη διακριτική ευχαίρεια του Συμβουλίου. Στην προηγούμενη ομιλία μου εγώ το χαρακτήρισα διευθυντήριο που κυβερνάει. Όχι, αυτό είναι λάθο τρόπο. Δεν μπορούμε από τη μια να διαδίδουμε τι κάναμε και να το προπαγανδίζουμε. Στη διεθνή πολιτική, στη διεθνή διπλωματία, ε, στο διεθνές εμπόριο χρειαζόμαστε μια ενιαία ευρωπαϊκή φωνή, μια ενιαία ευρωπαϊκή δράση, μια ενιαία ευρωπαϊκή στάση. Και ταυτόχρονα Όμω, λέει ο καθένα, ναι, αλλά μου ταιριάζει εθνικά αυτό. Αν δεν μου ταιριάζει, αν δεν είναι ευκαιριακό στην εσωτερική πολιτική, δεν το θέλω. Ε, όχι. Αυτό ακριβώ ε, συμβαίνει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να σας πω και κάτι, αυτό δεν χαρακτηρίζει ε, ειδικά μία κυβέρνηση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει τις περισσότερες κυβερνήσεις, αλλά έχουμε και εμείς σοσιαλιστικές κυβερνήσεις και σοσιαλδημοκρατικές. Όλες οι κυβερνήσει με τον ίδιο τρόπο αντιδρούν. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα, είναι θεσμικό. Και αυτή λοιπόν η θεσμική κατάσταση, ο θεσμικός κίνδυνος φέρνει σε κίνδυνο όλη την Ευρώπη. Και καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι, και αυτό είναι μια έκκληση τώρα προς όλες τις πολιτικές ομάδες, να πούμε όλοι ευρύτατα ότι αυτό που χαρακτήρισε ο κύριος Ντόλ κοινοτική μέθοδο να εφαρμοστεί. Γιατί ακριβώς είναι η εφαρμογή και η επιβολή των κοινοτικών αρμοδιοτήτων για τη λύση των προβλημάτων. Αυτό θέλουμε να γίνεται σε κοινοτικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ας πούμε έχουμε ένα νομισματικό πρόβλημα. Μπορεί ακόμα να λυθεί αυτό σε εθνικό επίπεδο. Ε, όχι. Μια οποιαδήποτε πρόκληση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να λυθεί σε, εθνικό επίπεδο. Όχι. Μπορεί οποιοδήποτε εμπορικό πρόβλημα στην παγκόσμια εμπορική πολιτική να λυθεί από ένα κράτος μέλος και μόνο. Και βέβαια με την Κίνα μπορούμε να ε, συνεργαζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε 500 εκατομμύρια και 27 εθνικές οικονομίες. Αλλιώ να διαλυθούμε στα εξώ συνετέθη. Μόνη της η Κύπρος, η Μάλτα, η Λετωνία, η Γερμανία, η Γαλλία. Γίνεται και αυτό. Δεν νομίζω ότι θα τους εντυπωσιάσουμε πάρα πολύ έτσι τους Κινέζους όταν θα πάτε να τους δείτε κύριε Βαν Ρομπέι. Γι' αυτό χρειάζεται η κοινοτική μέθοδος. Γι' αυτό είναι καθήκον του Κοινοβουλίου να επικρατήσει η κοινοτική μέθοδος και να την επιβάλλει το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά διαστόματος Μπαρόζο στα θέματα των Ρωμά ε, έδειξε ότι είναι έτοιμη να αγωνιστεί. Το θέμα των Ρωμά θα το λύσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να το λύσουμε. Και το Κοινοβούλιο θα το λύσει όπως είπαμε όλοι από κοινού. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Και αυτό ισχύει και για περίπλοκες μειονότητες. Γι' αυτό δεν θα ενδώσουμε εδώ. Αλλά κάποια στιγμή θα έχουμε άλλη πρόκληση στις δημοσιονομικές προοπτικές. Και τώρα σας προβλέπω ότι η στρατηγική επανεθνικοποίηση θα ξανάρθει αλλά θα προσκρούσει στη μαζική αντίσταση του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος... Ε, κύριε Σούλτς, κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Κύριε Σούλτς, συμφωνείτε για την ερώτηση. Η κυρία Μορβάη θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Είναι πολύ απλή ερώτησή μου, κύριε Σούλτς οι ιδέες των πολιτών στα κράτη-μέλη μας σε εσωτερικό επίπεδο. Πώς είναι δυνατόν να αγνοούνται πλήρως. Αυτό πώς εντάσσεται ε, στη γραμμή των βασικών ε, ελευθεριών και της δημοκρατίας. να λαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο αποφάσεις από μη εκλεγμένα πρόσωπα και αυτές να κυριαρχούν επί της ε, θέλησης των λαών των πολιτών. Πολύ απλή ερώτηση νομίζω. Ε, thank you, Mr. President Schultz. Ο κύριος Σούλτς, αγαπητοί συνάδελφε, κάθε κράτος δικαίου έχει το καθήκον να φροντίζει να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται το δίκαιο. Γι' αυτό συμφωνώ 100% με εκείνους που λέγουν ότι Εάν πρόκειται για μεμονωμένου πολίτε, ανεξαρτήτω προελεύσεω, ένα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί προκαλούν προβλήματα, είναι καθήκον του κράτου μέλου και των αρχών του να ε, λύσει τα προβλήματα. Α πούμε, αν είναι του ποινικού δικαίου να υπάρχει δίωξη. Αυτό ισχύει όμω αντίστροφα και για την επιβολή του κοινοτικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη που είναι κράτη δικαίου αλλά και είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση, είναι υποχρεωμένα να δέχονται και να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν και το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό απαιτούμε προκειμένου για τους Ρωμά τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκίφερ Χόφσταθ έχει το λόγο από του φιλελευθέρους και ε, δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Φαν για τις σημαντικές δηλώσεις ε, για το Συμβούλιο και θα ήθελα να αρχίσω με το τελευταίο μέρος ε, της παρέμβασής σας σχετικά με τους Ρωμά. Θα ήθελα να πω σαφώς και προσωπικά συνάδελφο του ΕΛΚ ότι σχετικά με το θέμα των Ρωμά η Κομισιό έδρασε με το σωστό τρόπο και δεν τους ε, δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε, πρέπει να τους βοηθήσουμε σε αυτόν τον αγώνα και θα ήθελα να κάνω έκκληση στην Επιτροπή να ε, μείνει ε, στη θέση της, διότι αυτό είναι ένα θεμελιώδες θέμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Νομίζω ότι οι αξίες είναι εξίσου σημαντικές όπως και οι κανόνες της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό όλοι να δουν ότι η Κομισιόν μεταχειρίζεται με ίσο τρόπο κάθε κράτος μέλος. Και τις μικρές χώρες και τις μεγάλες χώρες. Για τις αξίες δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα μικρά κράτη και στα μεγάλα κράτη. Πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Βεβαίως είναι αληθές ότι η Σύνοδος Κορυφής κατά κάποιο τρόπο καπηλεύθηκε από, από αυτό το θέμα Βεβαίως, πολύ συχνά ε, υπάρχει αυτό, διότι το θέμα της ημέρας καπηλεύεται τις εργασίες ενός ε, μια συνάντησης. Βεβαίως, δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο, δεν μπορούμε να ανεχθούμε να έχουμε μια νέα οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση ε, χωρίς αυτά τα νέα μέσα για την οικονομική διακυβέρνηση διότι ξέρουμε ότι ένας πυλώνας νομισματικός δεν μπορεί να σταθεί χωρίς έναν οικονομικό. Και αν δείτε τα spreads ανάμεσα στα επιτόκια τα γερμανικά και τα επιτόκια άλλων κρατών είναι πάρα πολύ ψηλά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα πακέτο υπεύθυνο επιτάπητος για την οικονομική διακυβέρνηση και ελπίζω ότι η Κομισιό θα έχει προτάσεις μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Για να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει το πακέτο αυτό να πληρεί κυρίως τρεις όρους. Ο πρώτος είναι, κύριε Πρόεδρε, όπως πάντοτε και εσείς είπατε, ότι δεν πρόκειται μόνο ε, για την δημοσιονομική εποπτεία, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε την μακροοικονομική εποπτεία. Και αυτό είναι το δίδαγμα από αυτήν την κρίση χρέους. Δεν είναι μόνο μια κρίση σταθερότητας, ε, ε, έχει επίσης και σχέση και με την κατάσταση της οικονομίας το πακέτο θα πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικές κυρώσεις και πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό είναι οι προοδευτικές κυρώσεις. Δεύτερον, ένα συντονισμό, έναν συνδυασμό οικονομικών ε, κυρώσεων και πολιτικών κυρώσεων. Όχι να υπάρχει επιλογή ανάμεσα στις μεν και στις δύο, να υπάρχει ένας συνδυασμός των δύο και τρίτον, σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξει αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου αυτών που παραβιάζουν τους κανόνες. Αυτό γίνεται στην κανονική ζωή, θα πρέπει να γίνεται και στην πολιτική ζωή. Και τρίτον, ο τρίτος όρος κατά το γνώμη μου κύριε Πρόεδρε είναι ότι θα πρέπει η Κομισιό ε, να ε, αρχίζει τις διαδικασίες αυτές, να ε, πυροδοτεί τις διαδικασίες, διότι άλλη εποπτεία δεν λειτουργεί, δεν λειτουργήσε με τη συνθήκη της Λισαβόνας, με το Σύμφωνο Σταθερότητας και δεν θα λειτουργήσει στο μέλλον. Είδαμε ότι το, η Γερμανία και η Γαλλία δεν τήρησαν στο παρελθόν το Σύμφωνο Σταθερότητας και άλλαξε. Πρέπει λοιπόν η ίδια η Κομισιό να ε, πυροδοτεί τις διαδικασίες και ελπίζω ότι στις 29 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τις προτάσεις και ε, θα έχουμε ένα αξιόπιστο πακέτο με βάση τις εργασίες της ομάδας δράσης ε, που θα μπορούμε να εξετάσουμε στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις παρατηρήσεις σας. Η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς, συμπρόεδρος των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Φαν Ρόμπαι ακούω την έκθεση πεπραγμένων για την τελευταία σύνοδο κορυφή που δεν πρέπει να τη λέμε λέτε σύνοδο, γιατί είναι απλώ συνάντηση του Συμβουλίου. Για τρίτη φορά ακούω αυτά που λέτε. Και οι δημόσιε δηλώσει μου προκαλούν σκέψεις και έχω την αίσθηση ότι εσείς και εμείς ζούμε σε άλλο γαλαξία. Τι περιμένω εγώ όταν συνεδριάζουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μαζί με υπουργού εξωτερικών στις Βρυξέλλες σε καιρούς οξύτατης κρίσης. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που μας παρουσίασαν. Όσο κηρύγματα και αν μας κάνετε για τη σύνοδο κορυφής που δεν επιτρέπεται να τη λέμε έτσι αλλά απλό συμβούλιο. Τίποτα δεν κάνανε τελικά. Και ειδικά ο δικός σας ρόλος κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου ως Πρόεδρου εκείνου που έκανε την ομάδα εργασίας, για την κρίση, για περισσότερη ε, οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Και ακριβώς το δικό σας ρόλο να το σκεφτείτε παρακαλώ. Χαίρομαι που άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνεχίζει αυτό το παιχνιδάκι που είναι προ όφελο του προσετερισμού περισσότερη ισχύω από τα κράτη-μέλη και θα κάνει προτάσει για το πώ ε, θα υπάρχει κοινή οικονομική διακυβέρνηση στι Βρυξέλλε. Έχω την εντύπωση ότι μεταξύ άλλων αυτή η αιμονή που έχετε ε, για την εστίαση και τη συγκέντρωση σε μηχανισμούς κυρώσεων, που έτσι κι αλλιώς δεν γίνονται χωρίς αλλαγή των συνθηκών, οδήγησε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Μια κατάσταση με τον μεταξύ των κρατών μελών που λέγουν ότι συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε. Αλλά πρόοδους για το στόχο που είναι περισσότερη οικονομική διακυβέρνηση δεν έχετε να ε, παρουσιάστε. Και παρακαλώ μην υποκρίνεστε εδώ όταν έρχεστε ότι δήθεν κάνουμε κάτι. Γιατί αυτό δεν βοηθάει σε περιπτώσεις τέτοιες, σε καιρούς κρίσης. Είναι πάρα πολύ ε, επιζήμιο εγώ βλέπω το ρόλο σας ε, ως ιδιαίτερη ευθύνη για προβολή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και έχω την εντύπωση ότι παρόλο που είναι δύσκολο αυτό το παιχνίδι των ρόλων ε, που σας επιφυλάσσει η συνθήκη της Λισαβόνας και οι αοριστείες της, θα πρέπει να φροντίσετε ε, να έχουμε πραγματική κοινοτική πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή δεν αντιποκρίνεστε στις απαιτήσει. Για τους Ρωμά πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ ότι ε, υπήρξε μονομερής ε, συγγνώμη από την κυρία Ρέντινγκ. Εγώ περιμένω να μας εξηγήσουν οι Γάλλοι γιατί σήμερα ανερυθρίασα ψεύδονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό δεν αξίζει καμία συγγνώμη. Ε, δεν το καταλαβαίνω. Χαίρομαι και για μένα είναι το καλύτερο συμπέρασμα της Συνόδου Κορυφής. Χαίρομαι που ο κύριος Μπαρόζο στήριξε την κυρία Ρέντινγκ. Αυτή η διαδικασία της προσφυγής στο δικαστήριο ε, για παραβίαση των συνθήκων πρέπει να ε, γίνει πραγματικότητα. Και με απασχολεί αυτό το γεγονός και η κυρία Ρέντινγκ έκανε αυτό το βήμα. Σε καιρού μεγάλη ανασφάλεια, οικονομική κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση, αβέβαιου μέλλοντο, ε, μεγάλη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αυξάνεται όλο και περισσότερο, με προβληματίζει αρχηγοί κρατών όπω ο Νικολά Σαρκοζή ή ο Σίλβιο Περλουσκόνη, πρωθυπουργό, θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλου, αλλά είναι οι πρωταγωνιστέ με το θεατρικό ε, όρο, με τη θεατρική έννοια του όρου τα πολιτικά τους προβλήματα και την αδυναμία τους ε, να κάνουν πολιτική, την ανικανότητά τους, την κρύβουν πίσω από τέτοια φαινόμενα. Σε αυτό το ρεπερτόριο που αγγίζει ε, την ξενοφοβία και τη μυσαλλοδοξία. Και θυμηθείτε τον περασμένο αιώνα εδώ στην Ευρώπη τι έγινε. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Κίρχοφ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Κύριε Πρόεδρε, Σύντομε παρατηρήσει πριν περάσω στην ε, βασική μου επισήμανση. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Συμβούλιο για το γεγονό ότι συγκεντρώθηκε στο θέμα τη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και έπειτα για του Ρωμά. Να καταστήσω σαφέ ότι ασκούμε ισχυρέ πιέσει για να γίνει σαφέ ότι θα ζητούσαμε μια νομική δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω θεματοφύλακα των συνδικών. Πρέπει να πω εδώ ότι το να κατηγορούμε μόνο τους Γάλλους ε, για κάποιες από τις κινήσεις τους στο επιτελείο τους δεν είναι πολύ επικοδομητικό ούτε σκόπιμο απόψη Ευρωπαϊκής ε, Ενότητας. Και για το Πακιστάν να πω ότι η χώρα αυτή είναι μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και είναι και μεγάλο εταίρος τουλάχιστον τριών ευρωπαϊκών χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν συμφώνησε για ένα συνολικό, μια συνολική δέσμη μέτρων όπου θα πρέπει να πληρούνται όμως κάποιοι όροι για να λαμβάνει αναπτυξιακή βοήθεια το Πακιστάν. Εδώ η αναπτυξιακή βοήθεια προς το Πακιστάν είναι ζωτική σημασία, Πρόεδρε, όπως και αλλού και η Βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει το ε, 5,7 του ΑΕΦ να το διαθέσει στο 2013 και εδώ πρέπει να πω ότι αυτό το σύστημα το στηρίζει μόνο, όχι μόνο η δική μας η ομάδα. Επίσης, κάθε ευρωπαϊκό έθνος σκοπεύει να δημιουργήσει μια ισχυρή εμπορευόμενη οικονομία. Το να βοηθήσουμε λοιπόν το Πακιστάν προς την πρόσβαση της αγορές με την άμεση άρση των ε, δασμών ε, για τις βασικές του εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό. Και παρόλο που βρίσκω λυπηρό ότι θα πρέπει να υπάρχουν χρονικά όρια σε αυτή την πολιτική, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατάσταση κατεύθυνση. Επίση, το να υπάρχει μια μεγάλη, μια σημαντική εταιρική σχέση στα εμπορικά ζητήματα Ευρωπαϊκή Ένωση και α, Πακιστάν είναι κάτι που και ο Βρετανό Υπουργό, ο κ. Κάμερον, το ανέφερε και κάτι που ο κύριος Ντέιβι, ο υπεύθυνο των εμπορικών συνομοσπονδιών στη χώρα μας, το υποστήριξε επίσης. Οι μηχανικές ανησυχίες που αναφέρονται στη δήλωση, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει τελικά από μια πρωτοπόρος πρωτοβουλία να μην γίνουν δειλά και ε, μέτρα χωρίς ε, τόλμη. Θα πρέπει εδώ, Πρόεδρε, να βεβαιωθούμε ότι όλες οι φιλοδοξίες της δήλωσης δεν θα δηληστούν από τους εγωιστικούς προστατευτισμούς. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Λεγιαρίκ από την Ενωμένη Αριστερά. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έδειξαν ότι οι διαξεφισμοί του Προέδρου της Γαλλίας και Τη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδήγησε σε ένα κυνήγι μαγισσών κατά ενό πληθυσμού της Ευρώπης. Το, ε, ε, στο όνομα της Οικουμενική δηλώση των ανθρώπων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η, Γαλλική, Αριστερά και άλλε παρατάξεις λένε ότι θα πρέπει αυτό αυτός ο διωγμό, ο επονίδητο διωγμό, να πάυσει. Και επίση θυμίζουμε και την οδηγία που ονομάζεται Επιστροφή του 2008, η οδηγία της ντροπή μιλά για την εταιρική σχέση η οποία απαγορεύει την απομάκρυση των Πακιστανών ε, χωρί ε, επαρκή δικαιολόγηση. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, κύριε Πρόεδρε, ώστε ο πληθυσμός των Ρωμά να βγει από την κατάσταση ένδυας και δυστυχίας στην οποία ζει. Η πολιτική κατά των μεταναστών ε, θα περιορίσει την ηθική και επιρροή που θα μπορούσε να έχει η Ευρώπη στον κόσμο. Και πρέπει εδώ να δούμε ότι ο λαϊκισμός κατά των μεταναστών ε, οδηγεί σε έξαρση του εθνικισμού και σε κάτι που είχε ονομάσει και ο Μπέρτορ Μπρέχτ ε, το επονίδι στο τέρας. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να θυμηθούμε ότι Πρέπει να είμαστε υπέρ των λαών και των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών. Να δώσω κάποια παράδειγμα. Τη στιγμή που ο φιλελευθερισμό οδηγεί τον κόσμο μα σε διεθνή κρίση, αναφέρατε εσεί στο κείμενό σα ότι θα πρέπει να έχουμε συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με πολλέ φιλοδοξίε. Μιλήσατε για επιτάχυνση τη διατλαντική αγορά και βεβαίω να συμμορφωθούμε προ του κανόνε των Ηνωμένων Πολιτειών και να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και στι δράσει του ΝΑΤΟ το να έχουμε φιλελευθερισμό στις αγορές, να υποταχθούμε στις ΗΠΑ και να στατικοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσουν σε αποτυχία. Μιλήσατε για σταδιακή κατεύθυνση σαφή τη Ευρωπαϊκής Ένωση, Μα τι εννοείται ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ενωμένη Αριστερά θεωρεί ότι η καλή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική δεν σημαίνει απλώ την καταπολέμηση τη ένδυα και τη φτώχεια, τον εκμηδενισμό των δανείων, την καταπολέμηση του υποσυτισμού, τον αφοπλισμό και την ειρήνη, αλλά ακόμη μια ενεργή πολιτική για να πετύχει και η Σύνοδο του Κανκούν για το κλίμα. Διότι το κείμενό σα λέει ότι είμαστε βεβαίω πρώτοι στι εμπορικέ συναλλαγέ, αλλά δεν σκοπεύουμε να φορολογήσουμε τι χρηματοπιστωτικέ ε, συναλλαγές επίσης. Ε, τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε στο το κείμενο αυτό να μας οδηγήσει σε έναν ισχυρότερο διάλογο, διαπραγματεύσει μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Ούτε στον ε, Ανατολική Ιερουσαλήμ ε, μιλάτε για πρωτεύουσα, στην αναφορά σας εκεί για πρωτεύουσα του Ισραήλ και ούτε είστε αυστηροί στις επικρίσεις σας προς το Ισραήλ. Και επίσης μιλάτε για σύνοδο ευρωπαϊκή και εποπτεία με ε, απειλή κυρώσεων κατά των κρατών μελών. Γιατί κρύβεται το γεγονός ότι τα κρατικά χρέη έχουν ε, ε, επιβαρυνθεί όχι μόνο λόγω των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και επειδή στηρίζονται μόνιμα τα, ε, οι δυνάμεις του κεφαλαίου. Ε, γιατί δεν στηρίζετε το βιομηχανικό και γεωργικό τομέα και δεν τον ξαναχτίζετε σε νέες βάσεις, γιατί δεν βρίσκεται νέους τρόπους να στηρίξετε την απασχόληση. Τι νομική μάχη σκοπεύετε να δώσετε για να επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση των κρατών και των λαών. Βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Έτος κατά της φτώχειας. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να αναλάβετε Ευχαριστώ κυρία Νίκη Τσαβέλα παρακαλώ, εξ ονόματος της ομάδας της. Κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των Ρωμά, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η απέλαση των Ρωμά από τη Γαλλία. Το πρόβλημα είναι οι απάνθρωπες ε, συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι Ρωμά στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και αντί να είμαστε καταγγελτικοί εδώ, θα έπρεπε όλοι μαζί να έρθουμε και να προτείνουμε εφόσον οι ρωμά είναι μια εθνική μειονότητα σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα να προτείνουμε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο ένα πανευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα για τους ρωμά στα πλαίσια του κοινωνικού αποκλεισμού. η απέλαση είναι μια παράμετρος του προβλήματος. οι συνθήκες που ζουν οι ρωμά είναι το πρόβλημα. κύριε πρόεδρε ως προς τα συμπεράσματα του συμβουλίου θέσατε τις εξωτερικές σχέσεις της ευρώπης μέσα στο πλαίσιο των αμοιβαίων συμφερόντων. αναμφίβολα η κίνα που διαθέτει 2,5 τρει εκατομμύρια δολάρια αποθεματικά και αναζητά να επενδύσει στην ευρώπη είναι μια πολύ συμφέρουσα συμμαχία. εν ώψη λοιπόν της ευρωκινεζικής συνόδου προτίθεστε να εξομαλύνετε τα εμπόδια που θέτει η ευρώπη στις σχέσεις της με την κίνα συγκεκριμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σχέσεις με το ιράν. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Φρανκ Φανέκε από τους μη Ευχαριστώ πρόεδρε. Η επίσημη ημερήσια διάταξη κανονικά της Συνόδου Κορυφής επισκιάστηκε πάρα πολύ από την πολιτική ορθότητα και την ανοησία τελικά και τις δηλώσεις κυρίας Ρέτινγκ κατά της γαλλικής πολιτικής ε, ε, για τους Ρωμά. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακληθεί στην τάξη. Έχουν δικαίωμα και όχι μόνο δικαίωμα τα κράτη-μέλη αλλά και καθήκον να αντιμετωπίζουν την απαράδεκτη επιβάρηση, ε, την ε, ένδυα των παιδιών, την παιδική ε, εργασία και τη λαθρομετανάστευση. Είναι υποχρεωμένα να προστατεύουν τους πολίτες τους. Και το να παραγνωρίζουμε τα προβλήματα των Ρωμά Τσιγκάνων δεν λύνει τίποτα. Θέλω να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνετε ένα καταβλισμό στον Περλεμόν μπροστά στην αυλή Ρωμά. Ο λεγόμενος πρόεδρος Βαν Ρομπέι και το Συμβούλιο και πάλι μια τρύπα στο νερό έκαναν. Μεγάλα λόγια, μεγαλώστομες δηλώσει, αλλά στη συζήτηση καμία σπονδυλική στήλη. Αυτά τα έχουμε συνηθίσει. Δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω ότι είναι περί... περίεργη αυτή η διαπίστωση ότι χάρη στην ιδιαίτερη στάση της Γαλλίας και της Ιταλίας, περασμένη φορά και πάλι αντιστάθηκαν ε, κάποιοι ε, στο πολιτικό πραξικόπημα των διορισμένων ε, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ήταν επιτυχία επιτέλους αυτό για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα θέλατε να πείτε, φαντάζομαι, λίγα λόγια για να δώσετε μια σύντομη απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μερικά λόγια για να απαντήσω σύντομα. Υπάρχουν πάντοτε διάφοροι τρόποι για να εκθέσει κανείς τα πράγματα. Μπορεί κανείς να οδηγηθεί από διάφορες αντιλήψεις, από τα επιτεύγματα και από τα γεγονότα. Ο χαρακτήρας μου τίνει μάλλον να με κάνει ε, να ακολουθώ την πραγματικότητα της επιτεύξης. Τι κάναμε κατά τη διάρκεια αυτών των οκτώ πρώτων μηνών του έτους με μια νέα επιτροπή και με νέα θεσμικά όργανα από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε για μια εποπτεία χρηματοπιστωτική σημαντική, μεταρρυθμίση εξαιρετικά σημαντική με τη συνεργασία βεβαίως του Κοινοβουλίου. Συμφωνήσαμε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις για μια δράση εξωτερική για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ένα νέο Υπουργείο Εξωτερικών, μια νέα διπλωματία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύο επιτεύγματα εξαιρετικά σημαντικά που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο μιας θεσμικής αρχιτεκτονικής περίπλοκης, αλλά την οποία θελήσαμε, επιδιώξαμε. Συμφωνήσαμε για ένα πακέτο σημαντικό για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να μπορέσει να επιβιώσει συμφωνήσαμε για ένα πακέτο 110 δισεκατομμυρίων με ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων εξαιρετικά σημαντικό επίσης και που πραγματοποιείται παρά τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες προσκρούει η ελληνική κυβέρνηση. Συμφωνήσαμε για ένα πακέτο 750 δισεκατομμυρίων στήριξης χρηματοοικονομικής στην περίπτωση όπου και βεβαίως υπό όρου στην περίπτωση όπου θα χρειαστούν πράγμα που καθησύχασε τις αγορές και δημιούργησε εκ νέου προοπτικές. Υπό την όθηση της Ένωσης, μεγάλες μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται και ξέρω ότι αμφισβητούνται βεβαίως μέσα στη χώρα και πέραν της χώρας. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χωρίς την πίεση που άσκησαν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης αυτό δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Στην εξωτερική πολιτική τώρα, θα το υπενθυμίσω, συμφωνήσαμε με 27 μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις κυρώσεις στο Ιράν για πρόσθετες κυρώσει εμείς, πράγμα που δεν ήταν προφανές εκ των προτέρων. Συμφωνήσαμε για ένα ψήφισμα με τους 27 σχετικά με τον διάλογο ανάμεσα στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πέντε, ακόμα πέντε χώρες ευρωπαϊκές δεν έχουν αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο. Αυτός ο διάλογος ενέχει μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή αυτή η οποία είναι επίσης μια ευρωπαϊκή ζώνη που θα πρέπει να έχει και μια προοπτική ευρωπαϊκή. Συμφωνήσαμε για μια εμπορική συμφωνία επιτέλους με την Κορέα. Συμφωνήσαμε για ένα πακέτο στήριξης όχι μόνο χρηματοοικονομικής αλλά και εμπορικής για το Πακιστάν. Συμφωνήσαμε για την συνολική προσέγγιση για τη Μέση Ανατολή και το Δεκέμβριο 2009 εκπονήσαμε μια κοινή θέση των 27 ε, σε μια από τις πιο αμφισβητούμενες περιοχές του κόσμου, τη Μέση Ανατολή. Και προσθέσαμε, προσθέσαμε μια νέα δήλωση την οποία επανέλαβε το κουαρτέτο πριν από μερικές μέρες. Όλα αυτά έγιναν, είναι επιτεύξεις όλες αυτές, είναι γεγονότα και εγώ εγώ προσπαθώ ε, να ακολουθώ τα γεγονότα, να μιλάω για τα γεγονότα, για την ομάδα δράσης τώρα. Εργαζόμαστε ε, βραδέως ίσως. Όχι, όχι. Αρχίσαμε το Μάιο και τώρα βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο. Είμαστε στο Σεπτέμβριο και σε μερικούς μήνες κάναμε μεγάλα βήματα πρόοδου και ε, θα καταλήξουμε όχι το Δεκέμβριο όπως προβλεπόταν, αλλά το, στο τέλος του Οκτωβρίου και σας διαβεβαιώνω ότι θα έρθω εδώ να αναφέρω τα ποιοτικά ε, πορίσματα που θα είναι σημαντικά της ειδική αυτής ομάδας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ανάμεσα σε εμά και την Κομισιό. Εργαζόμαστε μαζί, συμβαδίζουμε για να επιτύχουμε ε, καλά ε, αποτελέσματα. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα στα όργανα αυτά. Σχετικά με το πρόβλημα των ΡΟΜ, των Ρωμά, επαναλαμβάνω τα πέντε σημεία που ήταν όχι πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διότι δεν συμπεράναμε αλλά νομίζω ότι για αυτά τα πέντε σημεία υπάρχει μεγάλο κονσένσους. Τώρα περιμένουμε τις έρευνες που πραγματοποιεί η Επιτροπή. Δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουμε τα πράγματα και επισημαίνω, όπως μου είχε ζητηθεί στο Συμβούλιο Κορυφής, ότι η Κομισιόν άρχισε τις εργασίες της για ένα σχέδιο για μια καλύτερη ενσωμάτωση πολλών μειονοτήτων, εκ των οποίων και η Ρωμά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσθέσω ακόμα μερικά λόγια στα Ολλανδικά που είναι μια μειονοτική γλώσσα ίσως, αλλά από καιρού εις καιρόν πρέπει να ακούγεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι ο απολογισμό των πρώτων μηνών σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες παρά το πείσμα των καιρών ε, ε, ήταν θετικός. Ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα ανέκαμπτε τόσο γρήγορα η οικονομία. Μπορεί να είναι η ανάκαμψη εύθραυστη, μπορεί να είναι η αρχή ακόμα. Αλλά αν μας το είχαν πει αυτό πριν από λίγους μήνες, ότι σε μία χώρα η οικονομική ε, ανάπτυξη μεγέθυνση θα φτάνε στο 3,5% ή κατά μέσον όρο στην Ευρώπη περίπου 1,5% κανείς δεν θα το πίστευε πριν από μερικούς μήνες. Ουδή. Σε κάποιες χώρες σε πολύ εξαιρετικά δύσκολες ε, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες εφαρμόζονται μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, εργαζόμαστε για ένα νέο είδος οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Σήμερα η κατάσταση είναι, και το λέω με προσοχή, και στην οικονομία και στην αγορά εργασίας καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, πριν από λίγους μήνες. Και αυτό είναι τυχαίο. Δεν νομίζω. Έχει γίνει κοινή προσπάθεια και συγκροτημένη και συγκεκριμένη. Και ένα τελευταίο. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από εμά όχι μόνο σήμερα, μία αντιπαράθεση και ε, μία συζήτηση για το ποια μέθοδος είναι η ενδεδειγμένη, η καλύτερη. Και εγώ θεωρώ ότι η κοινοτική μέθοδος όντως, αλλά οι πολίτες περιμένουν κυρίως αποτελέσματα να τους δώσουμε και κυρίως μία προοπτική. Αν είναι καλύτερες οι προοπτικές, μπορούμε να το λέμε ανοιχτά και θα έχουμε μεγαλύτερο όφελος από την εμπιστοσύνη των πολιτών και από την υποστήριξή τους για την ευρωπαϊκή ιδέα. Λοιπόν, εγώ προσανατολίζομαι στα γεγονότα. Δεν ε, ε, αφήνω να με ε, κυβερνούν ε, κάποιες αισθήσει και εντυπωσει που έχω για την κατάσταση. Εγώ σας λέγω ότι έχουμε κάνει πρόοδους, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω θα τη διατηρήσουμε και να βελτιωθεί ακόμα η κατάσταση από ό,τι ήταν ε, πριν από μερικούς μήνες. Σας ευχαριστώ. Uh, Παρακαλώ, κύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, Κάποιε αντιδράσει σύντομε στι δηλώσει των αρχηγών των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα για το θέμα των Ρωμά. Και εδώ να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει τι δύο βασικέ της κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα ενδελεχή διεξοδική ανάλυση απονομική άποψης της όλης κατάστασης και έπειτα στήριξη προ του Ρωμά και την ένταξή του, Διότι γνωρίζετε ότι όλοι κάνουμε εκκλήσει και ζητάμε ευρωπαϊκέ λύσει εδώ και καιρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω έχει εργαστεί πολύ σκληρά σε συνεργασία με την Ισπανική Προεδρία προκειμένου να οργανώσει το σχετική σύνοδο στην Κόρδοβα. Και ξέρουμε ότι δεν ήταν τόσο υψηλή συμμετοχή. Πρέπει λοιπόν να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία, αυτή τη συζήτηση, να τη δούμε ω ευκαιρία για να ξαναρχίσουμε την εξετασία τη στρατηγική μα, να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε του πόρου και τα μέσα μα καλύτερα για το μέλλον. Διότι είναι σαφέ ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή συνένεση για τέτοιου είδου ζητήματα. Χρειαζόμαστε τη δέσμευση και τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των εθνικών αρχών και των αρχών τοπική αυτοδιοίκηση, τη κοινωνία των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τι δυνάμει μα προ μια κοινή κατεύθυνση και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε θετικές λύσεις για το πρόβλημα των Ρωμά στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Εδώ να διαβεβαιώσω τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων ότι οι προτάσεις μας πρόκειται να αντιμετωπίζουν ζητήματα μακροοικονομικών ε, προβλημάτων ισορροπίας μέσω της ε, εποπτείας. Θα ενισχύσουμε το προλογικό πλαίσιο και το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας ε, επικεντρωνόμενοι στην ε, βιωσιμότητα και τον περιορισμό των κρατικών ε, δανείων με λιγότερο παρεμβατισμό. Όλα αυτά θα προταθούν στις 29 Σεπτεμβρίου ένα πακέτο με πέντε προτάσεις κανονισμών και μία πρόταση οδηγίας. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες που έχουν αναφερθεί από τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων θα αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το πακέτο προτάσεων που θα υποβληθούν συντομότατα, όπως σας είπα. Σε ό,τι αφορά το Πακιστάν, νομίζω ότι ήδη έχουμε κάνει πολλά και παραμένουμε οι βασικοί ε, διεθνείς συνεισφέροντες ε, στο Πακιστάν και εκεί αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος μας. Όμω είμαστε ακόμη στα πρώτα βήματα για το πώ μπορούμε να βοηθήσουμε το Πακιστάν. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, πρέπει να είμαστε πιο συνεπεί στην προσέγγιση μα και πρέπει να συνδυάσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξιακή καθώς και με τη βελτίωση της πρόσβασης των ε, προϊόντων του Πακιστάν ε, στην εμπορική διάσταση, την αγορά της Ευρώπης. Αυτά πρέπει να γίνουν στο δυνατόν συντομότερα. Και για αυτό το λόγο πρέπει να συναβαδίζουμε με τους κανόνες του ΠΟΕ και με τους υπόλοιπους εμπορικούς μας εταίρους. Αλλά αναζητούμε συνεχώς τρόπους για το πώς να δημιουργήσουμε την ε, επιληξιμότητα του Πακιστάν για το GPS, ε, το GPSP για το 2014. Όσο για την Μέση Ανατολή, εδώ νομίζω ότι είναι γενικός παραδεκτός στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή ότι αυτή είναι μια από τις βασικότερες προτεραιότητές μας στο διεθνές προσκήνιο να σας διαβεβαιώσω ότι η Βαρονιάστον είναι πολύ ενεργή στην όλη διαδικασία και ήδη εξετάζει πώ μπορεί να συνεργαστούμε ε, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνουμε αυτέ τι ε, διαπραγματεύσει και είναι σε επαφή με όλου του ε, πολιτικού ευθύνοντε σε αυτή τη διαδικασία. Ο κ. Ντόλ είπε ότι η επιτάχυνση αυτή τη διαδικασία είναι σημαντική. Σα διαβεβαιώ ότι από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίω τη κυρία Άστον θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δραματίσουμε εδώ τον ζωτικό ρόλο που μα αρμόζει. Σα ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Άλλοι αγορητές. Κύριο Σίβο Μπελέτια, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε πάει καλημέρα σας. Σωστά σας άκουσα να λέτε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν αποτελέσματα από μας και προοπτική να τους δώσουμε. Και νομίζω ότι η πρώτη προϋπόθεση που πρέπει εμείς να τους έχουμε είναι να μιλούμε μία φωνή, ενιαία φωνή και ε, στη Σύνοδο Κορυφής επόμενες εβδομάδες με την Ασία και τον πρόεδρο Ομπάμα είναι η φωνή μα μία και θα εκτιμηθεί. Μία από τις βασικότερες προτεραιότητες των επομένων μηνών είναι η συζήτηση για το κλίμα, Πρόεδρε. Και ως Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω θα πρέπει να τολμήσουμε να καταθέσουμε νέες πρωτοβουλίες. Και εδώ σκέφτομαι το όλο θέμα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η λεγόμενη προσέγγιση ρομπέν των δασών. Ορίστε, ας είστε εσείς ο ρομπέν των δασών, ο νέος. Και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ε, στην εξοικονόμηση ενέργειας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρική. Γιατί και εσείς γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε ε, ότι έχουμε δεσμευτεί για στην Αφρική δραστικά να περιορίσουμε την ε, φτώχεια. Ε, να ποντάρουμε στην αηφόρο ε, ενέργεια και αυτό θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι αποτελεσματικό εργαλείο για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο και να μην αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο μόνο στους Ασιάτες, βλέπε Κινέζους στην Αφρική. Κύριε Φαν Ρόμπεϊ, τελειώνω. Ε, μέχρι τώρα ήταν άψογη η πορεία σας ε, μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν περίμεναν πολλά από εσά. Σα θεωρούσαν απολύτω άγνωστο. Τώρα προσβλέπουν όλοι σε εσά. Έχετε βάλει τα θεμέλια για καλά βήματα στο μέλλον και ε, την οικονομική και χρηματοπιστωτική θύελα καταιγίδα την έχουμε ξεπεράσει και μόνο ευκολότερα. Καλύτερε μέρε μα περιμένουν τώρα. Ευχαριστώ η κυρία Βερονίκ Ντεκεζέρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι ε, περιμένουμε από ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση οικονομική και ε, ε, μας ήρθαν οι Ρωμά. Περίμενα πολλά από την κυρία Ρέντινγκ, την υποστηρίζουμε και για την φόρμα και για την ουσία. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε ε, συνεχώς αναφερόμαστε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο διότι θα αντιλήσουμε κανένα δίδεγμα. Οι Αθήγανοι όπως και οι Εβραίοι όπως και οι ομοφιλόφιλοι όπως και οι κομμουνιστές πήγανε στα στρατόπεδα, εξολοθρεύτηκαν και η κυρία Ρέντινγκ έχει δίκιο όταν λέει ότι από τότε, από την εποχή εκείνη αποφασίσαμε και την Ευρώπη και την ειρήνη και να μην, υπάρχει, να μην υπάρχουν πλέον διακρίσεις ε, εναντίον ε, ενός φίλου, μιας φιλής ε, εμείς εκτιμούμε το πώς είναι θεματοφύλακας των συνθήκων και ε, εκτιμούμε και φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο και στα μεγάλα και στα μικρά κράτη και μετά από το Συμβούλιο αυτό βλέπουμε ε, την άνοδο νέων εθνικισμών κάτι που είναι για μένα μια εμπειρία τρομερή, τρομακτική που έχει ένα άρωμα της δεκαετίας του 30 που εμένει. Θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό για την οικονομική διακυβέρνηση. Πολύ σύντομα είπατε ότι η ομάδα δράσης προχωρά στη δουλειά της. Τον Οκτώβριο θα έχουμε συμπεράσματα. Θα έχετε μηχανισμούς εποπτείας με την πιο αυστηρή ορθοδοξία την οικονομική. Ναι, αλλά μας μιλάτε και για τα κοινωνικά θέματα, για τα συντάξεις, για τις κοινωνικές παραμέτρους. Πού είναι όλα αυτά. Λέτε ότι αυτό ε, είναι ευθύνη των κρατών. Όχι, αυτή δεν είναι η γνώμη της ομάδας μας. Θα πρέπει να υπάρξουν παράμετροι κοινωνικές. Δεν μπορούμε να οικοδομούμε την Ευρώπη ε, κατά των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάντηση εργασία ήταν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εξωτερική πολιτική αυτή και συνέπεσε περίπου ε, ε, τα Ηνωμένα Έθνη και την Κίνα και στη Γενική ε, Συνέλευση ψηφίστηκε η Καταψηφίστηκε μάλλον η δική σας αναβάθμιση και η αναβάθμιση της κυρίας ε, Άστον. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε με τους Κινέζους αυτά ε, στο μέλλον. Είναι μακρύς ο δρόμος προς την πολιτική ένωση, προς την πολιτική δύναμη. Σήμερα είμαστε οικονομική δύναμη, αλλά οι πολίτες περιμένουν να λύσουμε την οικονομική κρίση και να αποδείξουμε ότι είμαστε δύναμη. Για την ομάδα εργασίας Task Force, είπατε κύριε ε, Φαν Ρόμπαϊ ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση. Τέλη του μηνός θα το δούμε, αυτό θα δοκιμαστεί. Στις 29 Σεπτεμβρίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, καταθέσει τη δική της πρόταση. Εσείς είπατε ο ίδιος στις 27 θα κάνετε την πρότασή σας. Ελπίζω περίπου να τα έχετε συνεννοηθεί αυτά και να έχετε συντονίσει. Πολύ καλή η κοινοτική σας ε, προσέγγιση και μέθοδος και καλό που μιλήσατε και Ολλανδικά. Ε, ωραία που, αυτά που λέτε για τη συνένεση, για την υποπτία, Η δημοσιονομική πολιτική των κρατών επίσης να ελέγχεται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Για τις κυρώσεις λέτε χρειάζεται μεγαλύτερη δουλειά. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό διαφωνία στο Συμβούλιο. Λοιπόν, όλα αυτά θα δοκιμαστούν τέλη του μηνός. Γιατί επιμένουμε τόσο πολύ για την κοινοτική μέθοδο εμεί ω Κοινοβούλιο. Το είπε ο συνάδελφο Σούλτ. Ε, αρχίζουμε να ε, εφαρμόζουμε τώρα τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι, το Συμβούλιο είναι ε, θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό, το έχει καταλάβει το Συμβούλιο, γιατί καμιά φορά μα φαίνεται ω συνέλευση εθνικών συμφερόντων. Ένα σαφέστατο εθνικό συμφέρον είναι του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο γίνεται να μην ρυθμίζουμε τα οικονομικά. Μα η κοινοτική μέθοδο ε, είναι μοναδική ευκαιρία να επιβάλλουμε το κοινοτικό συνολικό συμφέρον επί των εθνικών συμφερόντων των μεμονωμένων. Γι' αυτό χαίρομαι που το είπατε με τόση ακρίβεια και στα Ολλανδικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζιλ Εύαν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι αποφασιστική στιγμή αυτή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ότι έχει ρόλο πρωταγωνιστικό διεθνώ, ιδίω στι κλιματικέ αλλαγέ και την καταπολέμηση τη φτώχεια, αλλά και την οικονομική διακυβέρνηση εσωτερικώ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, να δούμε το έλλειμμα διακυβέρνηση από τη συνθήκη τη Λισαβόνα και να έχουμε ολοκληρωμένε ευρωπαϊκέ προσεγγίσει. Να αναγνωρίσουμε τη σημασία της περιφέρεια, των περιφερειών ε, στην συνολική διακυβέρνηση και να επαναλάβουμε το στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Εδώ λοιπόν το, το, θα καλωσορίσω τον Πρόεδρο Μπαρόζο στην εκλογική περιφέρεια στην Ουαλία την ερχόμενη εβδομάδα. Και ελπίζω ότι θα μιλήσουμε για την καταπολέμηση των υψηλών επιπέδων που έχουμε εκεί φτώχεια, μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη. Θα δείξουμε πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφέλησε την οικονομία μα και τι κοινότητέ μα και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το είδου η πρόοδο ε, και σε άλλε περιοχέ ε, όπου δεν θέλουμε να υπάρχει εθνικοποίηση των πολιτικών μόνο από τα κράτη-μέλη και βεβαίω το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην θέσουν σε κίνδυνο τα ε, καλώ λειτουργώντα ευρωπαϊκά συστήματα για σκοπούς οικονομική και χρηστής διακυβέρνηση. Ευχαριστούμε. Ντύρκ Γιάννέπινγκ, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Φερχόφστατ να παραμείνει στην αίθουσα. Η Ρωμά είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρώπη ε, βαθιά ριζωμένο. Όχι τόσες υποκρισίες. Ακούσαμε τον κύριο Φερχόφστατ ε, στην προηγούμενη ε, σύνοδο να κατηγορεί τον κύριο Σαργοζή για πράγματα που έκανε ο ίδιος το 1999. Ο κύριος Φερχόφστατ απέλασε προς τη Σλοβακία Ρωμά. Ομαδικά. Και καταδικάστηκε το Βέλγιο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν. Γι' αυτό, κυρίε και κύριοι, το σώμα έχει δικαίωμα να γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολίτε. Γιατί το λέω αυτό, Διότι. Α, αυτό δεν με ακούει ο κύριο Φερχόφστατ. Κάνουμε διάφορε περίεργε δηλώσει και δεν θέλει να του το θυμίζουμε. Αυτό ακριβώ κάνω κι εγώ. Γιατί έχω εκλεγεί για να θυμίζω στον κύριο Φερχόφστατ τα πεπραγμένα του. Και αν, πάρει ποτέ ε, αν ε, μάλλον ποτέ υπάρξει Νόμπελ υποκρισίας, είμαι βέβαιος ότι θα το κερδίσει με μεγάλη διαφορά ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριο Μπορκέτσιο για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, Νόμπελ για υποκρισία θα έδινα και στην Επίτροπο Ρέντι, η οποία ξέχασε να μιλήσει από τη φάνηκε από τις εμπειρίες μας, το τι γίνεται και με τους Ρωμά στο μεγάλο βουκάτο του Λουξεμβούργου. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα απλώς με τους Ρωμά, αλλά ότι δεν προβλέπεται από το νόμο η δημιουργία τοπέδων συγκέντρωσης. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας καλημερίσω γιατί είναι και πρωί και να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που όπου τελικώς ένας επικεφαλής ε, κράτος και κυβέρνησης άκουσε να δίδονται καλά μαθήματα πατριωτισμού ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν επιτρέπει μέσω των επιτρόπων της να προσβάλλονται κράτη-μέλη, όπως η Γαλλία, η οποία ξέρουμε ότι είναι υπέρμαχος των ενιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όλα αυτά ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαιώματος ε, που διαθέτουν οι λαοί. Το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν μας οδηγεί σε φιλετικούς λαϊκισμούς, αλλά όπως μας θύμισε και ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. The next speaker, Daniel Van Stoep. Κύριος Ντανιέλ Βαντερ Στούπ από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από 15 μέρες εδώ το Κοινοβούλιο γελιοποιήθηκε με το ψήφισμά του που φόρτωνε τα πάντα στη Γαλλία και την καταδίκαζε εκ των προτέρων. Περίεργη κατάσταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, καθόταν ε, στη θέση του δικαστή. Και μετά έρχεται εκεί η Επίτροπος και συγκρίνει τι καταστάσει με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλο. Κάτι πάει στραβά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική καταδικάζουν αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων χωρίς να γνωρίζουν την κατάσταση. Θα πρέπει λίγο περισσότερο να ασχολούμαστε με τα νομικά και τα δημοκρατικά θέματα. Τα νομικά ζητήματα είναι κάτι που αφορά τα κράτη και τους πολίτες και τα θεσμικά θα πρέπει να, δούμε ποιος θα πρέπει να τα τηρεί. Ως θεματοφύλακας το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχουν και δικαστές και εθνικοί και κοινοτικοί. Ε, ε, ε θελοντικά έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί οι Ρώμα και πήραν και 300 ευρώ στην τσέπη ο καθένας. Γιατί ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το νομικό δεν είναι θέμα εκτοπισμού ή απελάσεων. Είναι ε, θέμα ε, φιλοξενίας. Μα ο καθένας αποφασίζει ποιος θα μπαίνει στο σπίτι του, μπορεί να του κλείσει και την πόρτα άμα θέλει. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με πολίτες της Ένωσης που έχουν στρεβλή συμπεριφορά σε άλλα κράτη της Ένωσης. Και η απάντηση είναι ότι όταν κάποιος είναι άνεργος και παίρνει επιδόματα και ε, παρανομή και όλα σε μια χώρα, να μπορεί να απελάβνεται, ναι. Και τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να προβαίνουν σε δράσει υπέρ των πολιτών, να του προστατεύουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Λάγκεν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θαυμάζω την αισιοδοξία σας που μας αναφέρετε για την ενδιάμεση έκθεση της Task Force. Θα δούμε στο τέλος τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μεν, αλλά σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, όπως εσύ και ο κύριος Μπαρόζο, προτρέχετε, γιατί είπατε ότι μαζικά ανέκαμψε η οικονομία. Για σίγα λίγο, στο βαθμό που οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι σε αυτή την ανάκαμψη, δεν θα έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Και καλό είναι που διαπιστώνεται μεν τις πρόοδους και όλοι μαζί από κοινού ελπίζουμε να γίνουν και πραγματικότητα. Αλλά αν είχε περάσει η άποψη της κυρίας Λαγκάρτ και οι συζητήσεις ακόμα κρατούν που έλεγε ότι η Γερμανία λέει... ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά τη εις βάρος των άλλων κρατών τη Ένωση, δεν θα υπήρχε αυτή η ανάπτυξη. χωρίς την ατμομηχανή θα υπήρχε τέτοια ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση. Και όποιο φρενάρει την ατμομηχανή ε, ε, θα φρενάρει και το τρένο και δεν θα φτάσει ποτέ στο στόχο του και στον προορισμό του. Δεν είπατε για το ε, υπερβολικό χρέος και την επίλυση του θέματος αυτού και ανήκει και αυτό στη συζήτηση. Και δεν αρκεί πιστεύω να βάλουμε ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο. Εντάξει, σωστό είναι και καλό και μπράβο που το επιβάλλατε, αλλά χωρίς πιο ενισχυμένο αυτοματισμό τι εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, όχι στους Υπουργούς Οικονομικών, στο ΕΚΟΦΗΝ, τα μέτρα του Συμφώνου σταθερότητα δεν πρόκειται να μπορέσουν να επιβληθούν και ποτέ δεν θα τα συζητήσουμε. Και για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, που είναι σημαντικό αυτό, θα πετύχει μόνο εφόσον, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ε, κρατήσει η κοινωτική μέθοδος με συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριο Χιούς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση η ομάδα μου υποστηρίζει τις προσπάθειες για καλύτερο συντονισμό αλλά έχουμε δισταγμούς και επιφυλάξεις ως προς την κατεύθυνση της Κομισιόν. Είναι μια προσέγγιση χωρίς ισορροπία που έχουμε τώρα εδώ και μια δεκαετία. Ίσως ε, θα, οι πιο καλές αγορές ε, με πιο ισορροπημένους προϋπολογισμούς ίσως να φέρουν περισσότερη οικονομική μεγέθυνση και ευημερία. Είναι πρέπει να έχουμε καλή ισορροπία ανάμεσα ε, σε στόχους ε, που ίσως έρχονται σε σύγκρουση. Αυτό αγνοείται. Τι προτείνεται για τους 24, ε, εκατομμύρια ανέργους στην Ευρώπη. Μείωση κοινωνικής προστασίας. Αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε οικονομική διακυβέρνηση με ένα μείγμα πολιτικής ισορροπημένο για τα δημοσιονομικά και μέτρα για την απασχόληση. Θα πρέπει να συμβαδίζουν οι δύο στόχοι. Η αναμόρφωση του συστήματος θα είναι μια χαμένη ευκαιρία αν ασχοληθούμε μόνο με τα δημοσιονομικά και τη μείωση του δημοσίου χρέους. Αυτή η στρατηγική θα είναι κακή τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής πλευράς. Σας, ε, συνάδελφε Χιούζ, μια ερώτηση σας απευθύνουμε. Ο κύριος Λάμπστορφ. Ναι, κύριε Χιούζ, Ήδη πάρα πολύ συχνά έχουμε συνεργαστεί ε, και εκτιμώ τη γνώμη σας σχετικά με τα πέτρα που πρέπει ε, να λάβουμε τώρα. Νομίζω ότι εσείς και η ομάδα σας ε, περνάτε δίπλα από το θέμα. Μήπως λόγω της υπερβολικής χρέωσης των υπερβολικών δαπανών έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κρίση. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει τώρα να θεσπίσουμε δημοσιονομικές πολιτικές υγιείς και να μειώσουμε το χρέος για να ξεφύγουμε από την κρίση. Μικρόφωνο, μικρόφωνο παρακαλώ. Ναι, ο Στίβεν Χιούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να, ε, σε ένα λεπτό να απαντήσω με επιχειρήματα περίπλοκα. Νομίζω ότι βεβαίω ότι τα δημόσια οικονομικά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά ο χρόνος και η μέθοδο είναι επίση κρίσιμα. Αν το κάνετε τόσο γρήγορα όσο προτείνεται για να φτάσουμε στο 3% το 2013, αυτό θα μπορούσε να εξαλείψει κάθε δυνατότητα ανάπτυξη, να οδηγήσει σε στασιμότητα και σε μακροπρόθεσμη ανεργία χρειαζόμαστε μια δυτή προσέγγιση, όχι μόνο την μείωση του ελλείμματος. Σας ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε τόσο θερμές συζητήσεις στην αίθουσα της Ολομέλειας. Ο κύριος Μάουρο, για να 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις ε, με κάθε ειλικρίνεια από πλευρά μου προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα με τη συλλογιστική ότι έχουμε την ε, έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εμένα με εξέπληξε το γεγονός ότι μεταξύ των διορισμών ε, της Προέδρου Άστον αναφέρθηκε και ένας Ολλανδός στην Νότια Αφρική, ένας Γάλλος στο Τσάτ και ένας Ισπανός στην Αργεντινή ενώ ένα Ιταλό μόνο στην Αλβανία. Όσοι βρισκόνται αριστερότερα από μένα δεν θα δυσκολευτούν να πούν ότι αυτοί οι διορισμοί προκύπτουν από μια νεοαπικιοκρατική νοοτροπία. Δεν είναι ευρωπαϊκή προσέγγιση εδώ τη υπηρεσία αυτή και το ερώτημά μου είναι ειλικρινέ. Ποιο θα είναι ο ρόλο τη Ευρώπη στο μέλλον. Ο ρόλο τη Ευρώπη θα είναι απλώ να περιορίζεται και να ε, ικανοποιεί τι περιφερειακέ πολιτικέ των διαφόρων κυβερνήσεων των κρατών μελών, διότι τότε θα πάνε όλα στραβά. Και έπειτα για το θέμα των Ρωμά. Να πω ότι για πολιτικού λόγου βεβαίω μπορεί να γίνονται επικριτικά σχόλια κατά τη μια ή τη άλλη κυβέρνηση για τι λύσει που προέκρινε. Όμω, ε, παραμένει ένα πρόβλημα που μα διαφεύγει. Είτε το θέλουμε είτε όχι, το να κοινοτικοποιήσουμε το ζήτημα των προβλημάτων των Ρωμά και των λύσεων πρέπει να εξευρεθούν στο θέμα τους και το να κοινοτικοποιούμε την προσπάθεια της Ευρώπης να αντιμετωπίσει προβλήματα μεταναστευτικών ροών που έρχονται από το νότιο μέρος του κόσμου είναι κάτι μάτιο. διότι αν δεν βρεθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα συνεχίσουμε να τρογόμαστε μεταξύ μας χωρίς να καταλαβαίνουμε σε τι καταστάσεις δυσαρέσκειας μπορεί να ζουν οι πολίτες μας. Σας ευχαριστούμε, συναδελφοί. Κυρία Μπερές, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, για την υπόθεση των Ρωμά, νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν στη φάση αυτή τη συζήτησή μα να θυμίσουμε το σύνθημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση μέσα στη διαφορετικότητα. Αυτό το σύνθημα θα πρέπει να ισχύει και για του Ρωμά ένωση στην διαφορετικότητα. Ας ε, σεβαστούμε λοιπόν τη διαφορετικότητα των Ρωμά και ας θυμηθούμε ποια είναι η στρατηγική που μόλις αποφασίσαμε. Η στρατηγική του 2020 ορίζει την καταπολέμηση της, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς λοιπόν ε, να αναζητούμε τώρα νέες στρατηγικές αφού τις έχουμε στα χέρια μας. Ας ε, πάρουμε τη στρατηγική που ήδη έχουμε και ας την πρικοδοτήσουμε με τα απαραίτητα κονδύλια και θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα στο θέμα της ένταξης των ρωμάτων για την οικονομική διακυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι όλοι μιλούν για μια μεγάλη επιτυχία που θα καθορίσει το ευρωπαϊκό εξάμεινο α είναι. Όμω, ω τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώ ποιο θα είναι ο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εάν μιλάμε εδώ απλώ για τη διοργάνωση συζητήσεων στην Ολομέλεια, όπω πολύ συχνά γίνονται, νομίζω ότι δεν θα έχουμε επιτελέσει το στόχο μα. Και έπειτα, ε, επιτρέψτε μου να σα επικαλεστώ, διότι όταν συναντήσατε του Υπουργού Περιβάλλοντο και Κοινωνικών Υποθέσεων, ακούσατε τι είχαν να σα πούν. Όμω, η οικονομική διακυβέρνηση που σήμερα θα στρέφει την πλάτη τη στον εσωτερικό στόχο τη απασχόληση δεν θα είναι στο ύψος των προκλήσεων που έχουμε θέσει τους εαυτούς μας. Και σε εσά υπολογίζουμε ώστε η οικονομική διακυβέρνηση να είναι ισόρροπη. Δηλαδή να λάβει απόψεις και την απασχόληση ως πρώτη προτεραιότητα. Σας ευχαριστούμε, ε, ε κύριο Σάριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την εξωτερική πολιτική που είπατε ότι ήταν ένα από τα βασικότερα ζητήματα τη ε, Συνόδου. Η εξωτερική πολιτική δεν θέλουμε να είναι απλώ αντιδραστική, αλλά να είναι διορατική, σφαιρική και να προλαμβάνει καταστάσει. Και επίση να θέτει μακροπρόθεσμου στόχου. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα νομίζω ότι αφήνει να έχουμε υπερβολικές φιλοδοξίες ενάν υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν συνοδευτεί από περισσότερη κοινή εξωτερική πολιτική. Θα είναι απλά ένα μέσο και όχι αυτός σκοπό. Εδώ χρειαζόμαστε πολιτική σύγκληση. Χρειάζεται να συγκλίνουν οι θέσεις των κρατών μελών μεταξύ τους χρειάζεται να έχει μεγαλύτερο ρόλο ο πρόεδρο του Συμβουλίου που συγκεντρώνει του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση στι θέσει των κρατών καθώ και του Ευρωκοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια. Διότι μόνο έτσι θα λειτουργήσει αυτό το νέο όργανο και χρειάζεται και περισσότερη αρμοδιότητα στην εξωτερική πολιτική και υπάρχουν πολλά περιθώρια για τι βελτιώσει. Μία αρμοδιότητα ε, σημαίνει και γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα για την Ευρώπη των 27. Όμω η αρμοδιότητα δεν μπορεί να είναι γεωγραφικά ουδέτερη Πρέπει να είμαστε πιο πρόσφοροι, πιο αποτελεσματικοί, πιο σκόπιμοι στην εξωτερική μα πολιτική προ όφελο των κατώμελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των στρατηγικού μα εταίρου. Πρέπει να ορίσουμε ποιοι είναι αυτοί, γιατί ο κατάλογο μα είναι ιδιαίτερα μακροσκελή. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένα σε αυτόν τον κατάλογο. Θα πρέπει λοιπόν να οριστεί με προσοχή μόνο οι σημαντικοί εταίροι και μόνο όσοι συγκλίνουν μαζί μας την πολιτική μας και συμμερίζονται μαζί μας τις ίδιες αξίες, έχουν τους, ε, τις ίδιες ανησυχίες για τα σταδιακά ζητήματα, μόνο αυτοί αξίζουν να, ονομα, να ονομάζονται ε, εταίροι στρατηγικής σημασίας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σασόλη για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, την ε, περασμένη εβδομάδα παρακολουθήσαμε ένα θέαμα που ήταν αρκετά ανησυχητικό. Διότι ο κύριο Σαρκοζή και ο κύριο Μπερλουσκόνη αμφισβήτησαν τι συνθήκε που έχουν υπογράψει οι χώρε του. Καταλάβαμε ότι ο Πρωθυπουργό τη Γαλλία και τη Ιταλία βρέθηκαν σε δύσκολη θέση στι χώρε του, διότι υπάρχει και η Επιτροπή η οποία υποκλήθηκε στι ε, επιθυμίε του και υπάρχουν επικριτικά σχόλια γιατί φάνηκε ότι από κάποιου επιτρόπου θέλησαν να αφαιρέσουν το δικαίωμα τη ελεύθερη έκφραση. Όπω έχουμε θυμίσει επανειλημμένω από το κοινό Κοινοβούλιο, οι Ρωμά είναι Ευρωπαίοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα. Τα ε, ευρωπαϊκά ε, όργανα δεν θα πρέπει να μας εμποδίζουν να ξεκινήσουμε διαδικασίες με παραβάση, διότι αλλιώς παραβαίνουμε τις αρχές της ίδιας της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και θα πρέπει να συμμεριζόμαστε τις στρατηγικές που ισχύουν για να ε, εξέλθουμε από την οικονομική κρίση. Εκφράστηκαν φωνέ κατά του λαϊκισμού, κύριε Πρόεδρε, που σκορπίζει στην Ευρώπη φόβους. Αυτό το κοινοβούλιο στρέφεται στην Προεδρία σας και την Επιτροπή που και ζητούν απάντηση με περισσότερη κοινωνική διάσταση και περισσότερη έμφαση στο ρόλο των πολιτών. Αυτό είναι η πρόκληση του ερχόμενου ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Φρανσίσκο Χωσέ Μπιγιάν Μον, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φοβάμαι Μάλλον χαίρομαι που ε, ασχολήθηκε με την εξωτερική δράση το Συμβούλιο. Νέο ο κόσμος, ε, πολλού πόλου έχουμε και οικονομικούς και πολιτικούς και είναι λίγοι οι πρωταγωνιστές, ενώ οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες. Καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να τις αντιμετωπίσει. Όπως είπε πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση παίζει ρόλο και το μέγεθος. Γι' αυτό ε, λυπάμαι την περασμένη εβδομάδα για την ψήφο ε, στον ΟΗΕ για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ανησυχεί αυτό που ψηφίστηκε. Στο μέλλον θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να ετοιμάζουμε τις συνόδους κορυφής ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και πώς ψήφισαν στις 14 του μηνός και τα διμερή και τα πολυμερή ζητήματα. Ε, θέλουμε να κυβερνήσουμε την παγκοσμιοποίηση και να ενισχύσουμε το G20. Η συνεννόηση με τις Ηνωμένε Πολιτείες είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε κοινέ αρχές και αξίες, πολλές. Ελπίζω για τις 20 Νοεμβρίου και είμαι σίγουρος ότι θα ετοιμάσουμε σωστά τη ε, σύνοδο. Ευρωπαϊκή εξωτερική δράση λοιπόν θα πρέπει να σημαίνει μεγαλύτερη συνέχεια και μεγαλύτερη συνοχή. Αλλά ε, μαζί με την ε, εσωτερική ισχύ της Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί και η συνεργασία των 27 και των σημαντικότερων κρατών. Είναι σημαντικό, είναι αναπόφευκτο, ο δρόμος θα είναι μακρύς και δύσκολος, θα πρέπει όμως να το κάνουμε. Στην Ευρώπη Ήδη ακούμε για κάποιες ε, φωνές που λέγουν ε, εποχή μετά τη δυτικοποίηση. Κοιτάξτε, τρέχετε πάρα πολύ και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι διερμηνείς για να σας αποδώσουν. Μην μιλάτε τόσο γρήγορα. Η κυρία Ζήτα Γκουρμάη. One minute, please, okay. Αγαπητοί ε, πρόεδρε και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν 296 ε, εκατομμύρια εδώ και έχουμε όλες τις δυνατότητες να είμαστε μεγάλη δύναμη όπως ήμασταν ε, στο οικονομικό και πολιτιστικό τομέα. Δεν έχουμε όμως εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες, είμαστε διαιρεμένοι, ελπίζω να έχουμε κοινή δράση. Δεν έχουμε μια κοινή φωνή και νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική, η πολιτική άμυνας και ασφάλειας δεν έχουν αναπτυχθεί όσο πρέπει. Μια κοινή φωνή σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ε, μεγαλύτερο συντονισμό πολιτικής, κοινές πολιτικής. Είναι στο επίκεντρο ε, της εθνικής πολιτικής όταν ε, πρέπει να ε, παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Γι' αυτό χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Πρόεδρου Βαν και ελπίζω το Συμβούλιο να συνεχίσει το συντονισμό, να τον εμβαθύνει. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το στόχο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ε, κυρία Λίβια Γιάροκα, 1,5. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω ε, την δήλωση του Πρωθυπουργού του Ούγκρου Ορμπάν για την ε, στρατηγική σχετικά με τους Ρωμά. Αυτό το κοινοβούλιο προσπαθεί να αναπτύξει ένα κοινό πρόγραμμα για την ενσωμάτωση των Ρωμά και μετά ελπίζω το Συμβούλιο θα υποστηρίξει Προεδρία για μια κοινή λύση για ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η βασική αιτία σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτιση των Ρωμά δεν είναι αιτία ρατσισμού, ξενοφοβία, αλλά υπάρχουν αλληλεξαρτήσει πολλών πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Και δεν θα πρέπει βάσει της εθνότητας αλλά βάσει των οικονομικών χαρακτηριστικών να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε την πτώχεια των Ρωμά και των μη Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική πρέπει να, είναι μια αλυσίδα συντονισμένη ε, μέτρων, αλλά βασίζονται σε αμφίσιμα, αμφίσιμους δείκτες. Ε, θα πρέπει να έχουμε πολυεπίπεδη ε, πολιτική και θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο ούτως ώστε να μειώσουμε την πτώχεια μεταξύ των γενεών και να μειώσουμε την υποανάπτυξη. Σας παρακαλώ να μιλάτε πολύ, πολύ πιο αργά. Δεν είναι δυνατόν να μεταφραστείτε μακροπρόθεσμα το θέμα της πτώχειας ε, είναι σημαντικό για την, αυριανό διαβατήριο ούτως ώστε ε, να πρέπει όλοι ενδιαφερόμενοι να μοιραστούν το βάρος ε, η ΜΚΟ, τα κράτη και η Ρωμά η η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει την ίδια πολιτική τη στιγμή που οι προκλήσεις είναι τόσο μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές και οι συνέπειες εκλογών είναι τόσο επικίνδυνες. Θα πρέπει θαραλέα να μεταμορφώσουμε όλη την προσέγγιση μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία μου. Ο κύριος Αντιπρόεδρος ε, της ομάδας και Γιάννη Σφόμποντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω πρώτα ένα λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπαρόσο και η κυρία Ρέντινγκ δέχτησαν επικρίσεις από πλευράς μου την περασμένη φορά για τη στάση τους στο θέμα το Ρωμά. Τώρα έρχομαι να τους ευχαριστήσω ε, εντάξει τα λόγια τους δεν τα είχαν πάντα ζυγίσει σε ζυγαριά ακριβίας, αλλά η κυρία Ρέντινγκ ε, ίσως παρασύρθηκε στην επιλογή ε, των λόγων της γιατί την έπνιγε η κατάσταση αυτή. Και προς τον κύριο Φανρόμπα ήθελα να πω Εκτιμώ την καλή σας θέληση. Τώρα λέτε ότι θέλετε να μιλάτε εξ ονόματος των 27 με τον Κινέζο ε, Πρωθυπουργό. Τι θα τους πείτε όμως, δεν τα είδα από τα πρακτικά ποια είναι η γραμμή μας η κοινή για την Κίνα. Μετά για τις στρατηγικές που λέτε, της εξωτερικής πολιτικής. Εδώ δεν αναφέρατε καν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην πω το Κοινοβούλιο αλλά στην ε, στρατηγική για το εξωτερικό εμπόριο χρειάζεστε το Κοινοβούλιο. Θα το συμπεριλάβετε στην εκπόνηση της στρατηγικής και αν ναι με ποιο τρόπο. Και ένα τελευταίο, αυτό που είπε τώρα ο Λάμπστορφ, δεν μπορούμε να καθίσουμε και να παραδεχτούμε αυτό που αποφάσισε ο ΙΕ. Να είμαστε εμείς οι πληρωτές δηλαδή, αλλά να μην έχουμε λόγο για τα όσα συμβαίνουν. Τι πήγε εκεί στραβά. Θα πρέπει να το εξτάσετε κι εσείς ε, ως Συμβούλιο με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να δικαιωθούμε και στον ΟΗΕ και να έχουμε δικαίωμα λόγω σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάν Μαρινέσκου για 1,5 λεπτό. Ε, Πρόεδρε, το Συμβούλιο ε, συζήτησε για τις εξωτερικέ σχέσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην ξεχνάμε όμω ότι για του πολίτε αυτό που περισσότερο είναι σημαντικό είναι η οικονομική τους κατάσταση. Εδώ λοιπόν ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μα για τη συμφωνία που πετύχαμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, όμω εάν δεν εξεύρουμε δυνατότητε επιβολή κυρώσεων, τότε δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Πρέπει να μπορούμε να επιβάλλουμε κοινώσει, αλλά όχι δύο φορέ να επιβαρύνονται οι πολίτε. Ε, μία φορά από την έλλειψη τη αποτελεσματικότητα και μία δεύτερη φορά από την μείωση τη ευρωπαϊκή στήριξη. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε μέτρα ώστε να προλαμβάνουμε τι δυσκολίε των πολιτών και να μην έχουμε περισσότερε αρνητικέ συνέπειε ό,τι αφορά του Ρωμά τώρα. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε οφείλουν να συμμορφώνονται με το δίκαιο και τους νόμους. Και όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να σέβονται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όσοι δεν τα σέβονται, είτε πολίτες είτε κράτη-μέλη, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Στην συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, θεωρώ ότι το να υποστούν τις κυρώσεις οι πολίτες, των οποίων τα 100 των οποίων τα κράτη-μέλη δεν επιλύουν τα προβλήματα του επί τη ουσία. Αυτό δεν είναι δίκαιο, διότι δεν μπορούμε μόνο με ευρωπαϊκό τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα το Ρώμα. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη προορισμού και διέλευση να προβλέψουν καταλόγου και μέτρα για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο χρειάζονται κοινά προγράμματα, ενιαία προγράμματα, πανομοιότυπα που να εφαρμόζονται συγχρόνω σε όλα τα κράτη-μέλη. Και επίση για την υλοποίηση τέτοιων ιδεών δεν θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερε ιδέε ή να καταβάλουμε περισσότερα κονδύλια, απλώ να έχουμε πολιτική βούληση. Ευχαριστώ η κυρία Κορίν Βόρτμαν Κόλ. Ένα μισή λεπτό κι εσείς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε πάει. εσείς είστε για ε, ε, περισσότερη δέσμευση ε, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να βγει από αυτή τη ζούγκλα των εθνικών συμφερόντων και των μεγάλων εθνικών κρατών. Αυτό μόνο θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Ε, εσείς εργάζεστε σκληρά για μεγαλύτερη οικονομική διακυβέρνηση και είστε και στον καλό δρόμο. Αλλά πέρσι τέτοιο καιρό θα ήταν αδιανόητο το Συμβούλιο από κοινού να υποστηρίξει ε, την Ευρώπη ε, για την ενίσχυση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να σας υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όταν θα ασκήσει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει. Είναι σημαντικό και θα πρέπει να είναι φιλόδοξα τα πράγματα. Όταν πρόκειται για τις κυρώσεις, και κάτι άλλο που θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό, όταν πρόκειται για το πώς τελικά το Συμβούλιο συμπεριφέρεται ε, ως προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εθνικά σχέδια. Όταν κάνει κάποια συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή θα είναι πρόθυμο το Συμβούλιο να τις εγκρίνει, όταν αυτές ας πούμε απευθύνονται και στο Λονδίνο και στο Παρίσι ακόμα και τότε, αυτό είναι το σημαντικό. Και εκεί είναι ε, το εμπόδιο, εκεί να βάγισε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζεται το Συμβούλιο και να προσανατολίζεται από την ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γκοζές, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ότι εφόσον πρόκειται για το θέμα των Ρωμά, οι θέσει είναι ισορροπημένε, λογικέ και στραμμένε προ το μέλλον για την επίλυση του προβλήματο τη ένδυα αυτών των πληθυσμών. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σα πω ότι εξετίμησα τον τρόπο με το οποίο παρουσιάσατε τα επιτεύγματα των οκτώ τελευταίων μηνών. Το κάνατε με με ακρίβεια και νομίζω ότι δεν λέμε αρκετά τα όσα κάνει η Ευρώπη, δεν το τονίζουμε αρκετά και δεν τονίζουμε αρκετά το ρόλο του Κοινοβουλίου. Μιλήσατε ε, για την εποπτεία αυτό έγινε επειδή το Κοινοβούλιο θέλησε όργανα με αρμοδιότητα πραγματικά ευρωπαϊκή που μπόρεσε να θεσπιστεί αυτή η εποπτεία επειδή όπως ξέρετε το Συμβούλιο Εκοφήν του Δεκεμβρίου 2009 είχε πολύ πιο περιορισμένη μετριοπαθή θέση ως προς το θέμα αυτό. Το G20 θα έχει με τη Γαλλία Ευρωπαϊκή Προεδρία θα πρέπει να μιλούμε περισσότερο και περισσότερο με μία φωνή και να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον. Βασιζόμαστε σε εσά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσάμπα Ταμπάιντι. Ένα λεπτό. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φαν Ρομπέι. Βεβαίω, πιστεύω ότι οι δραστηριότητε σα είναι εξαιρετικά σημαντικέ. Είστε συστηματικό ε, και έχετε συνέπεια στη δουλειά σα. Πρέπει να πείστε τα κράτη-μέλη ότι η Ρωμά πρέπει να έχουν μια μακροπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στρατηγική για να ενταχθούν, να ενσωματωθούν. Στην Ουγγαρία έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Χρειάζονται προθεσμίε χρηματοδότηση για μια τέτοια στρατηγική. Ο κύριος Χέσκοβιτ από την Κομισιόν και ο κύριος Μπούζεκ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, πρέπει να συνεργαστούν για να υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθηση ούτως ώστε τα κράτη-μέλη ε, να πληρούν ε, πλήρως τις προϋποθέσεις, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με μια στρατηγική υπέρ των Ρωμά που να προσδιορίζει πιο ρόλο, ποιο ρόλο πρέπει να παίξει το περιφερειακό επίπεδο, πού είναι οι αρμοδιότητες και ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Θα, και θα έχουμε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από μια τέτοια στρατηγική. Ευχαριστώ. Σαρλ Γκόρενς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Βαν Ρομπέι, ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο θέλετε να ε, την ενότητα την Ευρώπη σε Ευρώπη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά κατά τη γνώμη ο τρόπος με τον οποίο εκπροσωπούνται στο G20 τα κράτη-μέλη ε, δημιουργεί δύο κατηγορίες ευρωπαϊκών κρατών. Αυτοί που είναι μέλη και αυτοί που δεν είναι μέλη οι έχοντες και μη μη έχοντες. Είναι αντίθετο προς την ενότητα και την ισότητα, την καταστατική. Δεν είστε της γνώμης, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι ο καλύτερος τρόπος για συνοχή και συντονισμό της οικονομίας της Ευρωπαϊκής στα πλαίσια του G20 είναι η Ένωση να αντιπροσωπεύεται από τα όργανά της, δηλαδή την Κομισιόν και το Συμβούλιο και όχι από μερικά κράτη-μέλη. Εάν η απάντησή σας είναι ε, θετική, πρόκειται να κάνετε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μην σηκώνουν τις μπλε κάρτες. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Είναι ένα ερώτημα. Θα σας παρακαλώ να ε, σηκώνετε την λευκή κάρτα αν θέλετε να λάβετε μέρος στην διαδικασία Catch the Eye. Η μπλε κάρτα είναι κάτι διαφορετικό. Σας έχουμε όλους στον κατάλογο, 25 άτομα στον κατάλογο. Δεν νομίζω ότι θα είναι δυνατό να μιλήσετε όλοι. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι η κυρία Κατρίν Γκρίς. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Βαν Ρομπέι, θα σας, είμαι ευγνώμων που υπενθυμίσατε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξία πυλώνας, αλλά με τις ξενοφοβικές δράσεις της γαλλικής κυβέρνησης, υποσχέσεις ε, μιας μελλοντικής πολιτικής δεν είναι στο ύψος των ε, προσδοκιών μας. Κύριε Βαν Ρομπέι, περιμένουμε μια καταδίκη, μια καταδίκη χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. Περιμένουμε προτάσεις συγκεκριμένες, την υλοποίηση των στρατηγικών που ήδη έχουν αποφασιστεί, κονδύλια, την αξιολόγηση των κονδυλίων αυτών και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Εν κατακλείδη θέλω να αφαιρθώ στα δικαιώματα και καθήκοντα που ανέφερε ο κύριος Ντόλ για να του πω ούτω ώστε να γραφτούν παιδιά στο σχολείο θα πρέπει να υπάρχουν λεωφορεία σχολικά και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται χρήματα. Ε, για το θέμα των Ρωμά δεν χρειαζόμαστε μόνο λόγια, χρειαζόμαστε κυρίως μια βούληση πολιτική σαφή χωρίς καμία αμφισημία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιοτρόφσκι. Παρακαλώ, για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, ήθελα να θίξω ένα σημείο επί της ουσίας από την αμερική διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ιδιαίτερη προτεραιότητα που θέλει να δώσει στι εξωτερικέ υποθέσει, στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υπηρεσία εξωτερική δράση και τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Εδώ το θέμα που προέκυψε με του Ρωμά και την απέλασή του από κάποια κάτι μέλη ήταν απρόοπτο. Ε, αλλά συνάδηκε με μια άλλη μέρημνα που ήδη είχαμε πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, εξαιτία τη συνθήκη τη Λισαβόνα, τα κάτι μέλη όλο και περισσότερο θα πρέπει να εξετάζουν τα ε, εγχώρια προβλήματα των ε, μετακινήσεων σε κοινοτικό όμως επίπεδο. Οι οδηγίε θα καταρτιστούν και τα μέτρα που θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να ξεπερνούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει νέα όθηση στις διατλαντικέ σχέσεις. Ελπίζουμε λοιπόν ότι στη σύνοδο με τον πρόεδρο Ομπάμα η αντιαμερικανική φοβία της Ευρώπης θα αντικατασταθεί από την προτεραιότητα που θα δώσουμε στον πραγματισμό μας και τα συμφέροντά μας. Δηλαδή να αρθούν οι υποχρεώσεις ε, θεώρησης για όλα τα κρατη μέλη. Παόλο ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Φανρομπέη για τα αποτελέσματα αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ιδιαίτερως για την προσπάθεια που συστηματικά κάνει για να στηρίξει την πραγματική οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια προσπάθεια που το ΕΛΚ και οι Πορτογάλοι βουλευτές του ΕΛΚ στηρίζουν. Έπειτα, χωρί να μακρηγορήσω, ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι προσπάθειέ τη, που από αυτή την άποψη έδωσε όλη την απαιτούμενη στήριξη και έλαβε όλε τι απαραίτητε πρωτοβουλίε την ε, κατάρτιση τη στρατηγική οικονομική διακυβέρνηση και ήθελα να κάνω και μια σύντομη αναφορά για την υπηρεσία εξωτερική δράση και κυρίω ε, για το άνοιγμά μας προ Πακιστάν. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι με αυτή τη χώρα, διότι σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις μας θα πρέπει να προστατεύουν τις χώρες οι οποίες ε, ε, καλύπτουν τους εργαζομένους τους δεν επιτρέπουν την εργασία των παιδιών και καλύπτουν με, κοινωνικό, με κοινωνικά μέτρα τους εργαζομένους τους. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φλασίκο Παρένοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ήθελα να θίξω κι εγώ δύο ζητήματα, ιδιαίτερα σύντομα, γιατί τα συζητήσαμε και προ 15 μέρου στην ε, Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Πρώτα απ' όλα για το θέμα των Ρωμά. Είναι αρκετά παράδοξο ότι Ήδη οι συνάδελφοι που έχουν επισκεφθεί καταβλισμούς Ρωμά δεν έκαναν κανένα σχόλιο σήμερα. Κάποιοι δεν έχουν μεταβεί ποτέ ως εκεί, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τα σχόλια αυτών που πήγαν. Ε, εγώ άκουσα προσεκτικά τι είπαν η κυρία Ρέντινγκ και ο κύριος Μπαρόζο. Ελπίζω λοιπόν ότι και με τις δηλώσεις τους αυτές θα καταφέρουν με επιτυχία να βρουν λύσεις στο πρόβλημα των Ρωμά. Το επόμενο θέμα που ήθελα να θίξω είναι η οικονομική διακυβέρνηση και ο ρόλος εδώ των κρατών μελών. Δεν υπάρχει μόνο η πολιτική σκοπιά εδώ, ούτε η ισότιμη εφαρμογή των μέτρων για όλα τα κράτη-μέλη. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στην εκτέλεση του προπολογισμού. Δηλαδή, να είμαστε σφαιρικοί στην προσέγγιση μας στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, δουλεύει το μικρόφωνο, εντάξει. Ωραία. Estar em destaque as graves contradições εδώ υπάρχουν μεγάλε αντιφάσει και αντίξωε συνθήκε που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μεγάλη δύναμη τη ε, παγκοσμίω, ε, είναι υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμω κυβερνήσει όπω η Γαλλία ε, παρουσιάζουν ε, συμπεριφορέ απαράδεκτε και ξενοφοβικέ, ιδίω σε σχέση με του Αθήγανου. Εδώ λοιπόν δεν λαμβάνονται εγκαίρω μέτρα ε, για την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά περισσότερο για σκοπού κερδοσκοπία και συγκεκριμένα κράτη δεν καταφέρνουν να καλύψουν, τα, να ανταποκριθούν στα παράλογα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητα και με παράλογο τρόπο απελάβουν πολίτε οδηγώντα σε καταστροφικέ συνέπειε λόγω των φιλελεύθερων πολιτικών. Επίση η αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θύματα του Πακιστάν και η συνεργασία. Αυτά δεν θα πρέπει να γίνουν ει βάρο των ευαίσθητων βιομηχανιών των χωρών που ήδη αντιμετωπίζουν δυσχέρειε και υψηλά επίπεδα ανεργία. Όπω ε, βιομηχανική τομή στην Πορτογαλία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προωθήσουμε πολιτικέ και να δώσουμε προτεραιότητα στην καταπολέμηση τη φτώχεια. Να ασχοληθούμε την παραγωγή πλούτου, την κάλυψη των δικαιωμάτων, την κοινωνική πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιόρδαν Σισελή τελευταία όμως για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Φαν Ρόμποϊ. Θα Ευχαριστώ κύριε Φαν Ρόμποϊ γιατί ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο σημαντικότατες διεθνείς συνόδους τον Οκτώβριο για την Επικοινότητα στην Ιαπωνία και την επόμενη στη Σεούλ για τις κλιματικές αλλαγές. Όλα αυτά υπό την αγίδα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα πρέπει βεβαίω να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε στο διεθνές προσκήνιο να έχουμε μια ισχυρότερη παρουσία, διότι γνωρίζουμε τι έγινε όταν σε κάποιες περιπτώσεις ε, υποστηρίξαμε διαφορετικέ θέσει μεταξύ μα. Δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα από τι διαπραγματεύσει. Εδώ θέλω να ρωτήσω τι εννοεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν λέει ότι πρέπει να μιλάμε με μια φωνή. Ε, πρόκειται εδώ να δεσμευτεί το προ αυτό και το ίδιο και η αρχική κατόχη κυβερνήσεων. Okay. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήσασταν πολύ γενναιόδωρος απέναντί μου στο χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να αντιμετωπίσω τα τρία βασικά θέματα που συζητήθηκαν σήμερα. Πρώτον, βλέπουμε την ισχυρή υποστήριξη για τη νέα στρατηγική προσέγγιση προς τους βασικούς εταίρους μας. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το πλαίσιο της Λισαβόνας και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την θέση της Ένωσης και την προβολή της ευρωπαϊκής δύναμης στην εξωτερική πολιτική. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με καλύτερη χρήση των συνεργειών της εξωτερικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα να δουλέψουμε σε επίπεδο κρατών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να, μιλήσουμε, για να μιλούμε με μία φωνή σε κάθε θέση. Γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα την σπουδαιότητα που δίνει ο κ. Βαν στην αποδοχή και ενσωμάτωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο από τα θεσμικά όργανα αλλά και από τους ηγέτες της Ένωσης. Όταν μιλούμε με μία φωνή, όχι μόνο πολυμερός αλλά και διμερός θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κάποια, κάποιες ε, Παρατηρήσει για την οικονομική διακυβέρνηση. Και εδώ βλέπω ισχυρή υποστήριξη στο Κοινοβούλιο για να συνεχίσουμε την πίεση που έχει ξεκινήσει για τις αλλαγές από την Άνοιξη και μετά, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο καλύτερο σύστημα. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους βουλευτές ότι δεν θα έχουμε ε, μόνο μια κριτική προσέγγιση στα δημοσιονομικά ελλείμματα αλλά και στα θέματα του χρέους, την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση του χρέους στο μέλλον. Επίσης πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να συζητά τα θέματα αυτά κατ' έτος, διότι κάθε Ιανουάριο η Επιτροπή θα έρχεται με την ετήσια παρακολούθηση το, της οικονομικής κατάστασης της Ευρώπης κάθε χρόνο, δίνοντας την κατάσταση της οικονομίας στα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης και θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε μια διεξοδική συζήτηση για το θέμα αυτό στο ξεκίνημα κάθε έτους. Ταυτόχρονα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ξεχνούμε τη σπουδότητα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική της, τα εργαλεία της στρατηγικής 2020 ε, της Ένωσης, ούτως ώστε να βάλουμε την ευρωπαϊκή οικονομία σε νέους τροχούς, σε νέες βάσεις, να προωθήσουμε την έξυπνη, πλήρη ε, και πράσινη ευρωπαϊκή προσέγγιση στην οικονομία, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση, την καλύτερη εκπαίδευση, τις πολιτικές ναι, για νέους υψηλής ποιότητας και την μείωση βεβαίως της φτώχειας. Και γι' αυτό απαιτείται καλύτερη εποπτεία και έξυπνες ε, οικονομικές πολιτικές παράλληλα, διότι μόνο έτσι θα πετύχουμε τα αναγκαία αποτελέσματα. Η Επιτροπή, αν θέλει κάτι είναι η έξυπνη επινόηση της κατάστασης. Εξωτερική υπηρεσία, ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, εδώ είναι σαφές ότι η κυρία Ιβαρόνι ε, Άστον θέλει να κάνει μια επαγγελματική υπηρεσία εξωτερικής δράσης που θα αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες, την ευρωπαϊκή δύναμη και το ευρωπαϊκό τοπίο. Γι' αυτό το λόγο η εξισορρόπηση γεωγραφική σε θέματα φύλου και, και σε θέματα προέλευσης είναι βασικό κομμάτι της δημιουργίας ε, αυτής της νέας επαγγελματικής ε, δομής προσωπικού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης όπως συμφωνήθηκε και η κάθε Άστον ανέλαβε τη δέσμευση να ενημερώνει τακτικά σε ό,τι αφορά την πρόοδο της ε, σύστασης της υπηρεσίας αυτής και νομίζω ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην μεταβατική περίοδο μέχρι το 2013 αποκρίνεται στις παρούσες ανησυχίες που κατανοώ πλήρω. Τελευταία παρατήρηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλου σα για την αιμονή σας ε, στο σεβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για την, τον ενστερνισμό των ευρωπαϊκών αξιών και την δέσμευσή σας να αναζητήσετε καλύτερες, ε, καλύτερους τρόπους ένταξης των Ρωμά. Ε, πάνω από 17,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για μέτρα υπέρ των Ρωμά και άλλων ευάλωτων ομάδων από την Επιτροπή και 12 κράτη-μέλη, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Πρέπει ωστόσο να δούμε πώς χρησιμοποιούμε και άλλα μέσα και εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ζητώ λοιπόν τη χρησιμοποίηση των μέσων αυτών με αποτελεσματικότερο τρόπο, με καλύτερο τρόπο και πιστεύω ότι για κάτι τέτοιο θα χρειαστούμε ε, μια νέα φρέσκια αντίληψη του μέλλοντος και μαζί νομίζουμε αποτελέσματα, πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα από τους παρελθόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mr. Vice President of the... Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει το λόγο. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσοι παρενέβησαν στη συζήτηση. Είναι αρκετά δύσκολο ε, να απαντήσω. Φυσικά από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρουσιάσει κανείς μέσα σε ένα λεπτό όλες τις απόψεις. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις, παρά μόνο ε, για δύο σημαντικά κεφάλαια θέλω να κάνω σχόλια. Πρώτον, της εξωτερικής πολιτικής. Είναι ένας δρόμος μακρύς. Έχουμε δει τη μεγάλη δουλειά που έκανε ο κύριος Σολάνα. Το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά αυτό. Σας απαρίθμησα ακόμα και το τελευταίο διάστημα ποιες είναι οι κοινέ θέσεις που μπορέσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να διατυπώσουμε για, τον, για το Ιράν και για κάποια εμπορικά θέματα. Κάναμε επίσης ένα βήμα πρόοδου σε σχέση παραδείγματο χάρη με τη θέση της Ευρώπης για τους G20. Είναι η μεγαλύτερη ετήσια παγκόσμια συνάντηση η G20. Όταν πήγα ως Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επί ένα, εδώ και ένα χρόνο γινόντουσαν ε, χωριστές συναντήσεις των κρατών μελών που ήταν μέλη των G20 και η κοινή τους θέση ήταν δική τους. Και ζήτησα, απέτησα από εδώ και στο εξή να υπάρχει κοινή θέση των 27 ακόμα και αν δεν παρίστανται όλες οι χώρες τους G20. Ο κύριος Μπαρόζο και εγώ εκπροσωπούμε την Ένωση ως Ένωση. Έχουμε λοιπόν κοινή θέση, σας διαβεβαιώ. Στην διάσκεψη των G8 και των G20 τα κράτη-μέλη και οι εκπρόσωποι της Ένωσης στέλνουν το ίδιο μήνυμα υπάρχουν στιγμές που υπάρχουν θετικά στοιχεία. Υπάρχει και πρόοδος και θέλω να σας υπογραμμίσω ότι σε αυτό το επίπεδο έχει σημειωθεί πρόοδος και επαναλαμβάνω είναι η μεγαλύτερη διεθνής παγκόσμια συνάντηση η G20. Προβλήματα υπάρχουν ακόμα φυσικά εξακολουθούμε να ζούμε την τραυματική εμπειρία της Κοπενχάγης. Υπήρχε μια κοινή θέση για ένα κοινό μήνυμα, αλλά δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε ε, τη θέση μας να γίνει δεκτή από τους αρτό. Αποτέλεσμα είναι ότι όλοι χάσαμε. Όλοι. Γιατί ως αποτέλεσμα αυτό είναι τελείως ε, μη ικανοποιητικό επί διαφόρων θεμάτων επετέύθη πρόοδος, αλλά φυσικά πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο πολύ για να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μου έθεσαν το ερώτημα. Ποιο θα είναι το μήνυμά σας στην διάσκεψη κορφής με την Κίνα σας καλώ να μελετήσετε, όχι επιφανειακά να διαβάσετε, να μελετήσετε προσεκτικά αυτά που περιγράφηκαν στο συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φυσικά, στο, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν θα περιγράψουμε τη στρατηγική μας, τις ε, ισορροπίες που θα παρουσιάσουμε στους στρατηγικούς μας εταίρους όπως είναι οι Κινέζοι. Αν όμως διαβάσετε το κείμενο, θα συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν νέα σημεία στα οποία βάζουμε έμφαση και υπάρχει αυτή η έννοια της αμοιβαιότητας. Δηλαδή δεν αντιδρούμε μόνο εμείς στα μηνύματα των άλλων, αλλά απέναντι σε αρκετούς εταίρους έχουμε αρχίσει να υποβάλλουμε αιτήματα. Και αυτή η αντίληψη υπάρχει, αυτή η αμοιβαιότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται και ακόμα περισσότερο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας εμπλέκεται στις ε, ε, εμπορικές συμφωνίες. Είσαστε συνομοθέτες για τις διεθνείς συμφωνίες και τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Άρα και εδώ έχει σημειωθεί πρόοδος. Πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα. Για τη διάσκεψη κορφής με τον Αμερικανό πρόεδρο θα, την προετοιμάσουμε στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Θα δουλέψουμε περισσότερο στο μήνυμα που θα δώσουμε ο κύριος Μπαρόζο και εγώ στον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα συμφωνήσουμε έτσι ώστε να μιλήσουμε εκ μέρους της Ένωσης, εκ μέρους των 27. Και πάλι λοιπόν, βήμα προς βήμα, θα προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερη παρατήρηση. Αφορά την οικονομική πολιτική. Τα δύο αυτά χρόνια εφαρμόσαμε μια έξυπνη οικονομική πολιτική. Πολύ πιο έξυπνη από ό,τι παλαιότερα. Έχουμε χαραμίσει 10 χρόνια. Μπορέσαμε να, θα μπορούσαμε να κινηθούμε εγκαίρως στο δημοσιονομικό επίπεδο, στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Δεν το κάναμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Μετά την ε, χρηματοοικονομική κρίση τι κάναμε. Δεν μιλάω για τη διάσωση των τραπεζών κτλ. Αλλά ακολουθήσαμε μια εξαιρετικά επικίνδυνη επεκτατική πολιτική το 2008 και σε μεγάλο μέρος και το 2009. Μια επικίνδυνη πολιτική γιατί αυξήθηκαν τα ε, δημοσιονομικά ελλείμματα. Αλλά από τη στιγμή που επήλθε η, ανάπα, η ανάκαμψη και το πιστεύαμε από, θα γίνει αυτό από την αρχή του χρόνου, από τη στιγμή εκείνη ξεκινήσαμε μια πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης, μια βαθμιαία μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων. Όχι απότομη, αλλά βαθμία. Ε, βαθμιαία. Κάναμε όμως και μια πολιτική ελαφρώς επεκτατική. Επίση, ακολουθήσαμε μια έξυπνη νομισματική πολιτική. Πάντοτε είχε ρευστότητα οι αγορές, ώστε να μην επιστρέψουμε στην κατάσταση της δεκαετίας του 30 ήταν αρκετά χαμηλά τα επιτόκια βάσει της πολιτικής μας για να επέλθει η ανάκαμψη και να μην ε, πληγούν ε, οι προπολογισμοί από τα πολύ ψηλά επιτόκια. Έτσι λοιπόν στο δημοσιονομικό και νομισματικό επίπεδο ακολούθησε μια πολιτική βαθμιαία, σόφρονα και ευφύ. Για ποιο λόγο, όχι για να έχουμε την ικανοποίηση να έχουμε σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, όχι για την χαρά του να μειώσουμε το χρέος, αλλά για να υπάρξει μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, για να μπορέσει να αποδώσει η πολιτική απασχόλησης. Όλες αυτές οι προσπάθειες είναι στην υπηρεσία της απασχόλησης υπάρχει μια προσπάθεια κοινωνική συγκεκριμένα μια προσπάθεια που θέλουμε να αποδώσει. Είναι εργαλείο και ο στόχος μας φυσικά είναι η απασχόληση και η μείωση της ανεργίας. Και όπως μόλις ακούσατε από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, για να τα πλαισιώσουμε αυτά ακόμα περισσότερο με κοινωνική διάσταση, έχουμε ενσωματώσει στους στόχους του 2020 τον στόχο της καταπολέμησης της φτώχειας. Έχουμε επίσης συμπεριλάβει την εκπαιδευτική πολιτική και διατηρούμε την πολιτική συνοχής, τα διαρθρωτικά ταμεία και πιστεύω ότι αυτά θα μπουν στις δημοσιονομικές προοπτικές που θα εκπονηθούν έτσι ώστε να έχουμε μια ως το δυνατόν δικαιότερη κατανομή σε όλη την Ένωση. Έτσι, ο στόχος μας από όλε τις πλευρές είναι κυρίως, κυρίως κοινωνικός και όλα τα άλλα παραμένουν δευτερεύοντα. Θα ήθελα να σας το πω αυτό στο τέλος αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την αναφορά που κάνατε εκ μέρους ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προχωρούμε στην επόμενη σημαντική συζήτηση τώρα στο Κοινοβούλιο. Περιμένουμε και τα εξελίξεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Λίγος χρόνος δηλαδή μεταξύ του προηγούμενου και του επερχόμενου. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαναρόμπουρη. Ε, ε, Συνεχίζουμε Αφού έχουμε ολοκληρώσει το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη,